Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto do... Καλό απόγευμα. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την ακρόαση για την ε, κοινή γεωργική προοδηγή με ε, χρονικό ορίζοντα του 2020 και ε, ε, θέλω να χαιρετήσω τους ε, συνομιλητές μας οι οποίοι θα φέρουν την έμπειρη γνώμη τους στη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να χαιρετήσω τον κύριο Άλμπερ Ντές ε, την κυρία, τον κύριο Πάολο Μπρούνι, την κυρία Σαβίνα θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω τον πρόεδρο της ΕΛΟ, ε, επίσης τον Μισελ Ντόουερ, καθηγητή Μισελ Ντόουερ, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Υπέθρου και θα ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Χάρμ Σπάντ, ε, πρόεδρος της, ε, του Γεωργικού Ευρωπαϊκού και Γεωργικού Συνεταιρισμού. Είναι χαρά για όλους μας που σας έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας, σε αυτό το ημικύκλιο. Είναι πολύ σοβαρή συγκυρία. Ε, είμαστε στην ε, στα πρόθυρα της υποβολής της, της Έκθεση ιδίας πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου για την γεωργία προς το 2020. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντομία το πρόγραμμα. Καταρχάς θα ε, έχουμε μία ομάδα, μία, ένα κομμάτι της... Συνεδρίασή μα θα το αφιερώσουμε στις άμεσες πληρωμέ. Ένα δεύτερο κομμάτι στα μέτρα της αγοράς και στο το τρίτο αφορά την ε, ανάπτυξη τη υπαίθρου έχουμε τις ερωτήσεις, ένα σχέδιο των ερωτήσεων που θα υποβληθούν και στο τέλος ε, θα έχουμε και μία παρέμβαση των μελών. Πριν, στο τέλος κάθε τμήματο, αν θέλετε, ε, αφού ολοκληρωθεί η παρέμβαση των, των, εισηγητών, θα σας ε, δώσω το χρόνο να, κάνετε, να γίνει μία σειρά ερωταπαντήσεων. Επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα στη διάθεσή μας, στο πρόγραμμά μας και να δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή μας ε, ταυτόχρονα, θα σας παρακαλέσω να σεβαστείτε το χρόνο σας, γιατί θα κλείνει το μικρόφωνο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Άλμπερ Ντέσσα, ο οποίος έχει 10 λεπτά για να μας παρουσιάσει το θέμα της ακρόασης. Έχει το λόγο, αγαπητέ Άλμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, σας χαιρετίζω και εγώ θέρμα και σας καλωσορίζω στην σημερινή ακρόαση για την αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2013 και χαίρομαι γιατί έχουμε εδώ εμπειρογνώμονες αξιούς και ε, προσβλέπω σε αυτά που θα μας πούνε. Σαν εισηγητής χαίρομαι πολύ για αυτή την ακρόαση. Είναι μία απόφαση της Δημοκρατίας δημοσία συζητήσεων και ε, τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν ή στην, εισαγωγή, ή στην εισήγησή μου. Θα μιλήσουμε για τις ε, τρεις πτυχές της κοινή γεωργικής πολιτικής, τις άμεσες πληρωμές, τα μέτρα για την αγορά και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Θα απογοητεύσω όσου νόμιζαν ότι θα παρουσιάσω σήμερα την εισήγησή μου, αλλά εάν ήταν έτοιμη η εισήγησή μου δεν θα χρειαζόταν η σημερινή ακρόαση. Ο Επίτροπος και τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, ζητούν ε, μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική σε μια διτή δομή βάσει των δύο πυλώνων. Οπότε πρέπει να αναπτύξουμε τη γεωργική πολιτική, να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει παραγωγή ποιοτικών τροφίμων και ε, αυτά πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μία αξιοποίηση των φυσικών πόρων αναφέρεται και στο εργατικό δυναμικό και στην βιοποικιλότητα για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι χώροι της υπαίθρου στα διάφορα κράτη. Ένας άλλος βασικός στόχος ο οποίος αναφέρεται στη στρατηγική του 2020 κατοπτρίζεται και εδώ. Πρέπει να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί η ύπεθρος και ε, ελπίζω ότι η ακρόασή μας θα συμβάλλει σε αυτό το με τα πορίσματά της. Εχθές στη συζήτηση ακούσαμε ότι ήδη στον αγροτικό χώρο της Ευρώπης ε, υπάρχουν περισσότερα απασχολούμενοι από όλη στην αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης. Είναι μία από τις ε, πιο βιώσιμες ε, γεωργίες ε, διεθνώς η ευρωπαϊκή και θέλουμε να βελτιώσουμε αυτή τη βιωσιμότητα με νέα μέτρα ε, για να υπάρχει μία αποτελεσματική ανάπτυξη και θα υπάρξουν διάφορα σχόλια γι' αυτό και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω όπου θα, θα καταλήξουμε σήμερα μετά από την ακρόαση για να υπάρχει μία ευρία εφαρμογή των σχολείων αυτών στην εισήγησή μου που θα ενσωματωθούν και υπάρχουν οικολογικά μέτρα για το περιβάλλον και αυτά μπορούν να αναπτυχθούν στο δεύτερο πυλώνα. Το ερώτημα είναι βέβαια πώς θα αναπτυχθεί ολόκληρο το σύστημα. Αλλά το προσόν των ε, οικολογικών μέτρων στον δεύτερο πυλώνα αιτιολογείται διότι τα μέσα θα πρέπει να ε, είναι μακροπρόθεσμα ενώ στον πρώτο πυλώνα θα ήταν μονοετή. Ε, πρέπει όμως να διαχωρίσουμε σαφώς τα μέτρα του πρώτου πυλώνα από αυτά του δευτέρου και αυτό θεωρώ ότι είναι για τη γεωργική πολιτική ένα πολύ βασικό θέμα ε, και γι' αυτό έχω στηριχτεί από πολλούς συνομιλητές μου όταν λέω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη είναι διαφορετικού μεγέθους. Γι' αυτό και κάθε ε, κράτος θα πρέπει ε, να προβλέπει ένα ποσοστό του ε, προϋπολογισμού για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ε, τώρα, όσον αφορά τον ορισμό των μικρών επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη, στα 27 κράτη-μέλη της Ευρώπης, θα πρέπει αυτό ε, να αφαιθεί στη διάκριση των κρατών μελών. Διότι άλλος θα αναφερθεί σε μία έκταση εκμεταλλεύσεως από, 200, από 2.000 τετραγωνικά, ενώ άλλοι θα μιλούν για 15 εκτάρια. Δεν μπορούμε εμείς να προδιαγράψουμε πώς θα αποφασίσουμε αποφασίζουν τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Αυτά θα χρειαστεί να αποφασίσουν, αλλά ήδη με ενδιαφέρει ότι θα πρέπει κάθε κράτος να χρησιμοποιήσει έναν ορισμό και να διαθέσει ένα ποσό για τους μικρούς αγρότες. Ε, ε, όσον αφορά τον ορισμό ε, των ενεργών γεωργών όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση του Επιτρόπου Τσόλος θα θέλω επίσης να αναφερθώ διότι θα πρέπει να υπάρξει μία αναδιάρθρωση των αμέσων πληρωμών προβλέπονται διάφορα πρότυπα αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούν να παραμείνουν οι μεγάλες διαφορές οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή με μαζί μεγάλων χωρών και χωρών σαν τη Λετωνία και άλλων. Άπαξ όμως και έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και ενημερώθηκα για τις μεγάλες διαφορές πρέπει να διαπιστώσω ότι υπάρχουν εξίσου μεγάλες διαφορές στις πληρωμές στο εσωτερικό των κρατών μελών. Υπάρχουν ορισμένα κράτη όπου οι γεωργοί ε, πληρώνουν, πληρώνονται μεταξύ 5 και 500 ευρώ ανά εκτάριο και σε άλλα κράτη ε, μιλάμε για διαφορά και διακύμανση από 50 μέχρι 500 στην ε, Ευρώπη και μεταξύ των κρατών μελών δεν πρέπει να υπάρχουν σημαντικές διαφορές και ακόμη λιγότερο τεράστιες διαφορές εντός των κρατών μελών. Αυτά τα θέματα πρέπει να λυθούν και γι' αυτό θα διατυπώσω προτάσεις όσον αφορά τις ε, διακυμάνσεις ε, των τιμών τις οποίες θέλουμε να αποφύγουμε θα πρέπει να διατηρηθούν τα ισχύοντα μέτρα για να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας σε περίπτωση μεγάλων αυξήσεων των τιμών των προϊόντων και θα πρέπει επίσης να αναφέρω ότι πολλοί συνάδελφοι μου είπαν ότι πρέπει να υπάρξει μία μεταρρύθμιση η οποία θα μειώσει την γραφειοκρατία και δεν θα την αυξήσει και ε, ε, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν θέλουν πλέον να ακούνε τη λέξη γραφειοκρατία διότι είμαι 20 χρόνια βουλευτής, 20 χρόνια μιλάμε για τη γραφειοκρατία και αντί να μειώνεται αυξάνεται. Σε αυτή λοιπόν τη γεωργική μεταρρύθμιση δεν πρέπει να συμβεί κάτι παρεμφερές και γι' αυτό όπως σας είπα εφόσον είμαι ευρωβουλευτής εδώ και 20 χρόνια ανέλαβε την επιχείρηση ο γιος μου αλλά μου είπε ότι εσύ πρέπει να συμπληρώνεις τις αιτήσει για να δεις τι αποφασίζεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Και είχε δίκιο, δεν φανταζόμαστε τι έχουμε αποφασίσει διαμέσου των ετών. Πρέπει λοιπόν να μειωθεί η γραφειοκρατία στη γεωργική πολιτική και να υπάρξει μία απλοποίηση των ε, κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης. Ε, επίσης αυτό θα πρέπει να ε, ισχύσει ε, για να μπορέσουμε μετά από το 2013 να έχουμε μία ισχυρή βάση χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Γεωργία για να υπάρχει παρκής δυνατότητα καλύψεως ε, και χρηματοδοτήσεως των εκτάσεων στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες έχουμε λάβει ορισμένες αποφάσεις, έχουν υπάρξει ορισμένες ψηφοφορίες όσον αφορά την ε, πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης. Χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι στο Στρασβούργο ψηφίστηκε με πλειοψηφίο δύο τρίτων τα πρότυπα τα οποία ζητούμε για τους Ευρωπαίους γεωργούς για την προστασία των ζώων, του περιβάλλοντος και των εδαφών να ισχύσουν και για το εξωτερικό. Και αυτό που θα με ενδιέφερε θα ήταν να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες που νομίζετε ότι πρέπει να εντάξουμε την συνιστόσα του περιβάλλοντα στον πρώτο πυλώνα ή στο δεύτερο. Πιστεύετε ότι η συνιστόσα θα πρέπει να συνδυαστεί με τις άμεσες πληρωμές. Τι θα γίνει με τις περιβαλλοντολογικές επιταγές. Πιστεύετε ότι χρειάζεται ένα ή περισσότερα προγράμματα. Σας ευχαριστώ εκ προημίου για τις απαντήσεις που θα μου δώσετε και σας ευχαριστώ ευχαριστώ γενικώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Άλμπερτο. Και τώρα ξεκινάει η συζήτησή μας με την πρώτη συνεδρία που αφορά τις άμεσες πληρωμές. Θα σας διαβάσω τον κατάλογο των πέντε ερωτήσεων και θα ήθελα να ζητήσω από το, ε, από το πάνελ να απαντήσει. Καταρχάς η πρώτη ερώτηση. Πώς οι άμεσες πληρωμές μπορούν να κατανεμηθούν ε, ισότιμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στους ε, γεωργούς. Δεύτερον, πώς ε, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΚΑΠ μπορούν να βελτιωθούν. Και εάν γίνει μια εισαγωγή μια, ενός πράσι, μιας πράσινης συνιστώσας, ποιο θα πρέπει να είναι το βασικό στοιχείο αυτής της συνιστώσας. Θα πρέπει, τρίτη ερώτηση, θα πρέπει οι άμεσες πληρωμές ε, να έχουν ένα ανώτατο όριο και αν συμφωνήσουμε πάνω σε αυτή την αρχή, ποια θα είναι τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν ε, στην, ε, στον περιορισμό αυτό. Τέσσερα, ποια, θα είναι, ποια είναι τα συγκεκριμένα, ποιο είναι το συγκεκριμένο σύστημα υποστήριξης για τους μικρούς παραγωγούς και πώς, και πώς μπορούμε να το ορίσουμε αυτό. Πέμπτη ερώτηση. Θα πρέπει μόνο η ενεργή παραγωγή να εισπράττουν τις άμεσες πληρωμές και αν ναι, πώς θα πρέπει να οριστεί αυτός ο ε, δραστήριος παραγωγός. Ας ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΚΟΠΑ να απαντήσει σε αυτές τις ε, πέντε ερωτήσεις μέσα σε οκτώ λεπτά, το μέγιστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε σε, αυτό το, σε αυτή την ακρόαση είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της ΚΑΠ και για όλους, και για τους παραγωγούς αλλά και για τους καταναλωτές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καταναλωτές ε, προφανώς είναι και αυτοί ε, έχουν αποφεληθεί από την κοινή γεωργική πολιτική, διότι αλλιώς χωρίς την ε, ΚΑΠ δεν θα είχαμε ε, τα, τα τρόφιμα τόσο καλής ποιότητας. Τώρα, για, το, για, την, για την πρώτη ερώτηση, πώς μπορεί να γίνει καλύτερη και πιο ισότιμη η χορήγηση των άμεσων πληρωμών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάποιες κάποια μέτρα τα οποία έχουν υιοθετήσει τα κάποια μέτρα, το ανέφερε και ο Αλμπερδές προηγουμένως, ε, θα πρέπει όμως να περιορίσουμε το γραφειοκρατικό σύστημα πληρωμών κάπως και η απλότητα, αν θέλετε, η απλούστευση θα πρέπει να είναι ένα ε, στοιχείο οποιοδήποτε μελλοντικού συστήματος. Ε, θα πρέπει να είναι απλό και από, από, από την πλευρά των υπηρεσιών αλλά και από πλευρά των γεωργικών Τώρα πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό το σύστημα. Νομίζω ότι μπορεί. Τώρα, το πρασίνισμα, αν θέλετε, της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής, ε, αυτό ίσχυε ανέκαθεν ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε μέτρα για την προστασία των ε, ε, των υδάτων επιφανείας, ε, τα είχαμε προστασία από τα ζωτούχα, ε, προστασία των βιοτόπων και του οικοσυστήματος γενικότερα. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα λαμβάνουν υπόψη του η παραγωγή. Μετά είχαμε και την γεωργία περιβαλλοντικών κριτηρίων για την υποστήριξη των γεωργών και ίσχυε ούτω ή άλλω ε, και ο κανόνα τη πολλαπλή συμμόρφωση. Οι παραγωγοί έπρεπε να προστατεύσουν ε, ε, του βιοτόπου, το φυσικό περιβάλλον κτλ. Ε, επίσης ο, ο αριθμός των ιζανιοκτώνων, των παρασιτοκτώνων που χρησιμοποιούνται ε, στην κοινότητα πρέπει να περιοριστεί. Βέβαια πολλά παρασιτοκτώνα χρησιμοποιούνται και στα εισαγόμενα, αλλά ούτως ή άλλως θα πρέπει τα ίδια, τα ίδια πρότυπα να χρησιμοποιούνται, ε, να επιβάλλονται και στα εισαγόμενα και στα εγχώρια προϊόντα. Επίσης θα πρέπει να υιοθετηθούν και άλλα μέτρα για την ειχνηλασιμότητα και η πρότασή της, στην πρότασή της η Κομισιό ε, συμπεριλαμβάνει μια σειρά μέτρων για το πρασίνισμα της κάπα Στο όμως τα πράγματα δεν είναι και τα ίδια όπως και στο παρελθόν, διότι ε, δεν είχαμε αλλαγή του κλίματος στο παρελθόν, ε, δεν είχαμε πρόβλημα με την παραγωγή των τροφίμων. Ε, τώρα πρέπει να διατηρήσουμε την ικανότητα παραγωγής μας. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε σταθερές τιμέ και σε άφθονη προμήθεια τροφίμων. Η ύπαρξη τροφή δεν πρέπει να θεωρείται σαν δεδομένο πλέον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλοντας μια πράσινη πολιτική υποβάλλει σε, ένα μεγάλο, ε, σε μια μεγάλη πίεση τους παραγωγούς της. Μερκασούρ, το, το Μερκοσούρ, το, Μαρό, το, Μαρόκο, η Βραζιλία, η Αργεντινή ε, έχουν συνάψει συμφωνίες ε, ε, ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν ε, κάνουμε και άλλες παραχωρήσεις σε αυτούς τους εταίρους μας θα αντιμετωπίσουν προβλήματα η παραγωγή μας. Δεν εξαρτώμεθα τόσο πολύ στις, στο γεωργικό τομέα από τις εισαγωγές όπως ας πούμε στον ενεργειακό τομέα. Επίσης θα πρέπει τα μέτρα τα οποία θετούνται να μην υποσκάπτουν την ανταγωνιστική μας θέση. Εάν μπορούμε να πετύχουμε ε, περισσότερο πρα, πρασίνισμα ας πούμε, μέσω της καινοτομία, τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, κανένα πρόβλημα. Αλλιώς ε, θα επιβάλλουμε άλλο ένα κόστος στους παραγωγούς. Κάτι το οποίο θα δυσκολεύσει, τους δυσκολέψει όσον αφορά την ανταγωνιστική τους θέση. Τώρα για το κατά πόσο πρέπει να πάει ένα το όριο για, την, για τις άμεσες πληρωμές. Εμείς δεν θεωρούμε ότι πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τέτοιου είδους ε, όρια, αν θέλετε, ανώτατα όρια, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε όλε, όλες αυτές τις υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ίχνηλασιμότητα, την ποιότητα κτλ. και ε, να παράγουμε όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται εάν ε, έχουμε τέτοιου είδους περιορισμούς. δεν ε, μπορούμε να εξαρτώμεθα μόνο από την αγορά. Και εφόσον όλοι η ενεργοί παραγωγή συνεισφέρουν στην ε, παροχή αυτών των ε, πλεονεκτημάτων για τους καταναλωτές, τότε όλοι θα πρέπει, όλοι οι ενεργοί παραγωγή να υποφελούνται οι ανισότητε που υπάρχουν ενδεχόμενα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα κράτη-μέλη μέσω τη φορολογική πολιτική. Η κοινωνική αγρογική κάπου δεν είναι μια κοινωνική πολιτική ούτω ή άλλω. Για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, συγκεκριμένο σχήμα υποστήριξη για του μικρούς παραγωγούς και πώ μπορούμε να το καθορίσουμε, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει, τι εννοεί η Κομισιόν μικρού παραγωγή. Οι περισσότεροι παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρή σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας σε άλλα σημεία του κόσμου. Το 80% των παραγωγών στην κοινότητα είναι κάτω από 10, ε, ε, ε, εκτάρια. Θέλουμε αυτές οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις να έχουν ένα μέλλον. Θέλουν όμως να γίνουν ταυτόχρονα και περισσότερες βιώσιμες μέσω βελτιώσεων στις υποδομές. Και αυτό θα γίνει μέσω της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η ανακοίνωση τώρα για τους, ε, μάλλον ο ορισμός των ε, ενεργών ε, παραγωγών. Το εξετάζουμε το θέμα. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Βλέπουμε την, στην Κομισιόν στην ανακοίνωσή τη λέει ότι οι πληρωμέ θα γίνουν στου ενεργού παραγωγού. Εμεί το εξετάζουμε στην κόπα αυτή τη στιγμή. Και ένα κριτήριο το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα είναι η σημασία του εισοδήματος που προέρχεται από τις γεωργικές δραστηριότητες σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το υπολογίσουμε και να το μελετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε για την ε, δυνατότητα που μας δώσατε και είμαι στη διάστηση για περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο τη ε, της ΚΟΠΑ, τον κύριο Walsh και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Ζαβίνη από την Βία Καμπεσίνα. Έχετε το λόγο. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα πολύ εύστοχα ερωτήματα μας ε, έδωσαν τη δυνατότητα να σκεφτούμε πιο συγκεκριμένα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως θα πρέπει να τα θέσουμε αντίστροφα βέβαια τα ερωτήματα αυτά, δηλαδή σε σχέση με την σημασία που έχει η διακύμανση των τιμών, η αστάθεια των αγορών και η ανάγκη παρέμβασης, ίσως καταρχάς πάνω σε αυτή την πτυχή. Πρόκειται για μια πρόταση την οποία στηρίζουμε με ε, έναν συνασπισμό οργανώσεων που προτείνει μια τέταρτη επιλογή, ένα τέταρτο σενάριο. Δηλαδή καθαρά ρύθμιση ε, των αγορών ώστε πρώτα να δούμε την, ε, πώς μπορούν οι τιμές να περάσουν ε, τα εισοδήματα και μετά να περάσουμε στις ενισχύσεις. Αυτό κυκλοφορεί γενικώ στους διαδρόμου, ως επιλογή τώρα. Σε ό,τι αφορά τις άμεσες πληρωμές θα θέσω λίγο αντίστροφα κι εγώ ε, για μια δεύτερη φορά το ερώτημα σε σχέση με τα 5-7 ερωτήματα τα οποία τίθενται. Πρώτα απ' όλα, είμαστε σύμφωνοι με τους στόχους της Κομισιόν για διατήρηση παραγωγής ε, τροφίμων σε όλη την κοινοτική επικράτεια να ε, λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τα εδαφικά ζητήματα. Η διατήρηση τώρα της παραγωγής τρομφίμων είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα σοβαρό θέμα σήμερα όταν λόγω των οικονομικών ε, δυσχεριών πολλοί αγρότες εγκαταλείπουν ε, το επάγγελμα αυτό. Μία έκθεση του Κοινοβουλίου φαίνεται να προβλέπει ότι ακόμα 4 εκ των 11 εκατομμυρίων αγρότες θα εξαφανιστούν. Είναι δύσκολη η δουλειά που έχουμε να κάνουμε και θα πρέπει να προσανατολιστούμε στον ενεργό δυναμικό, ε, στους ενεργούς αγρότες και να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους γεωργικούς παραγωγούς στην Ένωση για τα επόμενα χρόνια. Και εδώ τίθεται και το θέμα του ορισμού. Τι θα πει ενεργός αγρότης. Για μας είναι ένας αγρότης ο οποίος ε, κάνει τη δουλειά του παραγωγή τροφίμων, συμβάλλει στην παραγωγή τροφίμων, στην ασφάλεια τροφίμων στην Ευρώπη. Η δραστηριότητα οι πολλαπλές δραστηριότητες και η μερική απασχόληση μπορεί να αναγνωριστεί επίσης σε αυτό το πλαίσιο. Και υπάρχουν και σε όλες τις χώρες τρόποι αξιολόγηση τη ε, της δουλειάς που παράγει ο κάθε εργαζόμενος και έτσι μπορεί να αξιολογηθεί και η βάση ε, που θα χρησιμοποιηθεί για την ε, άμεσες πληρωμές, για την καταβολή της βοήθειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, νομίζω ότι έχει τεθεί, έχει λυθεί το ζήτημα, δεν χρειάζεται για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να γίνει μια ξεχωριστή κατηγορία γίνεται, ε, λαμβάνονται υπόψη με τις, ε, και οι μη αγρότες αν θέλετε ε, λαμβάνονται υπόψη στην κατηγορία. Δεν χρειάζεται μια ειδική κατηγορία. Τώρα σε ό,τι αφορά τους πρώτους εργαζόμενους μιας εκμετάλλευσης. Ίσως αν δοθεί εκεί προτεραιότητα θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ουσιαστική για τους μικρούς αγρότες. Πάντως σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο οι πιο μικρές δομές να ληφθούν υπόψη για την συμβολή που έχουν σήμερα στην ασφάλεια των τροφίμων και όχι για υποθετικές διαφορετικές ε, εξελίξεις ή διαφοροποίησεις. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ε, να πούμε ξεκάθαρο ότι είμαστε υπέρ του πλαφών στις πληρωμές. Κυρίως όμως να υπάρξει καλύτερη κατανομή σε όλους τους αγρότες και σε όλες τις χώρες. Θα δώσω ένα στοιχείο, ε, μην το γράψετε όμως, 100.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αγροτών, διαβάθμιση δηλαδή ανάλογα με τον αριθμό των αγροτών. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως να υπάρχει ένα αριθμητικό στοιχείο, ένα νούμερο, γιατί αυτό θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στον ε, γεωργικό πληθυσμό, ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει Ευρώπη πολλούς γεωργούς, πολλούς αγρότες και πρέπει να παραμείνει ζωντανή η πέθρος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επανεξισορρόπηση μεταξύ των χωρών, για μας η βοήθεια που δίνεται στο εργατικό δυναμικό, το γεωρικό, θα πρέπει ίσω να διαβαθμίσετε με βάση το μέσο εισόδημα ή το κατώτατο εισόδημα στη χώρα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει αυτή η η διαβάθμιση, η διαμόρφωση να χρησιμοποιηθεί για να τιμωρήσει εντό εισαγωγικών τι φτωχότερε χώρε που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. Θα πρέπει αυτή η διαβάθμιση να μπορεί αντίθετα να ενθαρρύνει την αύξηση του εισοδήματο και του γεωργικού εισοδήματο. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουμε αυτή τη διαβάθμιση των ενισχύσεων και με βάση την οικολογική συμμετοχή, τα οικολογικά αποτελέσματα. Από τον πρώτο πυλώνα λοιπόν είμαστε υπέρ. Από την πρώτη στιγμή υπέρ της ενθάρρυνσης, της παρότρινσης οι αγρότες να θετήσουν πιο οικολογικές πρακτικές και να παίρνουν κάποιες πρημοδοτήσεις για να χρησιμοποιούν τα πιο ορθά συστήματα να εφαρμόζουν συστήματα τα οποία καταπολεμούν πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι υπέρ της βιοπικιλότητας κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζουμε ότι η μια καθαρή στήριξη της βιολογικής οργανικής γεωργίας είναι απαραίτητη. Και επίσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν και βελτιωμένα συστήματα εκμετάλλευσης που λαμβάνουν υπόψη στο περιβάλλον. Μεταξύ αυτών, το θέμα των πρωτεϊνών νομίζουμε ότι είναι πρωταρχική σημασία. Πρέπει να ευνοήσουμε την παραγωγή των πρωτεϊνών στην Ευρώπη. Αυτό έχει ευεργετικά ωφέλη και για το περιβάλλον, μικρότερη ανάγκη να έχουν αυτά ζωτούχα λοιπάσματα και καλύτερη συμβολή στην ε, προστασία του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι με αυτό πανόραμα το σκιαγράφησα και το χρόνο μου τήρησα και απάντησα στα πέντε ερωτήματα που είχα στο χαρτί που έχω μπροστά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σαβίνη. Τον λόγο έχει ο πρέσβης κύριος Κοράντο Πίρτσιο Μπυρόλη. Για την πρώτη ερώτηση σχετικά αφορά τις άμεσες πληρωμές. Ήθελα να πω ότι εμείς σαν ΕΛΟ συμφωνούμε με τις άμεσες πληρωμές όσον αφορά ε, για, την, ε, για τις άμεσες πληρωμές. Θα πρέπει να πληρώνονται βέβαια με βάση τα εκτάρια και σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν ορίσει τα κράτη-μέλη. Οποιαδήποτε και αν είναι τα κριτήρια βέβαια τα οποία αποφασίζονται φασιστούν, οι πληρωμές ούτως ή άλλως ε, θα, είναι, θα γίνουν δύσκολες. Βέβαια, καλό θα είναι να μην, γίνονται, να μην γίνεται πληρωμή κατά με, με, με μέσους όρους, αλλά να έχουμε ανώτατο ή κατώτερη πληρωμή. Λοιπόν, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι οι πληρωμές αυτές ε, θα γίνονται με βάση την επιφάνεια, τότε πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα απλουστευτεί το, απλουστευτεί το σύστημα. Επίσης, ε, ένα χαρακτηριστικό των άμεσων πληρωμών είναι η σταθερότητα του εισοδήματος. Κάτι το οποίο επιτρέπει στους παραγωγούς να αντισταθμίσουν την διακύμανση και τους κινδύνους διακύμανσης ε, του εισοδήματός τους. Όσον αφορά την ε, περιβαλλοντική επίδοση, το πράσινο δηλαδή, θα πρέπει να δώσουμε μια μεγαλύτερη ε, όθηση στο πρασίνισμα της ΚΑΠ. Ε, αυτό θα γίνει μέσω των διαφόρων πυλώνων, δεν πρόκειται να πω σε λεπτομέρειες, αλλά περισσότερα δημόσια αγαθά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εκτό από τα μέτρα του άρθρου 68, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είμαι θα αντί, αντίθετη στην ιδέα τη Κομισιόν να εισάγουμε ε, ε, πρασίνισμα του, του πυλώνα 1 σε συνδυασμό με την πολλαπλή συμμόρφωση. Πιστεύουμε ότι αυτά μπορεί να γίνουν καλύτερα μέσω πολιετών συμβολέων και θα έχουμε καλύτερη και πιο έγκαιρη ε, υποβολή δημόσιων αγαθών μέσα στα πλαίσια του πυλώνα 1. Και, αλλά όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει μια κατανομή ανάμεσα στους δύο πυλώνες, διότι θα επικρατήσει μια σύγχυση. ensure... Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι η προσπάθεια των κρατών μελών και των μεμονωμένων παραγωγών ε, έχει, δεν πρέπει να ε, τεθεί σε κίνδυνο. Ερώτηση 3 όσον αφορά τα ανώτατα όρια. Όχι, όχι, όχι, δεν πρέπει να υπάρχουν. Λόγω, ε, για λόγους αρχής και πρακτικούς λόγους. Ούτως ή άλλως, ε, ο ορισμός ορίων θα πλήξει περισσότερο τις ε, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αν θέλετε, και τις πιο πράσινες εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη και θα περιορίσει και την ανταγωνιστικότητα. Αυτό θα γίνει αν εισάγουμε ανώτατα όρια. Η εμπειρία στις Ηνωμένε Πολιτείες δείχνει ότι ε, θα υπάρχει μια κούρσα ανάμεσα στους ε, εκμεταλλευτές, στους, ε, στους ιδιοκτήτες των εκμεταλλεύσεων για να δούνε ποιος είναι αυτός ο οποίος δικαιούται περισσότερο, ποιος έχει παράγει τα καλύτερα, ποιος δικαιούται να πάρει εκείνο κτλ. πιστεύω ότι θα ήταν ε, θα ήταν πολύ, θα ήταν πολύ καλύτερο να έχουμε μια καταποκοπή πληρωμή ανάλογα με την επιφάνεια των ε, εκμεταλλεύσεων. Οι περισσότεροι όμως παραγωγοί που δικαιούνται κάτι τέτοιο ε, αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα. Εξού και δεν χρειάζεται να έχουμε ιδιαίτερες, ιδιαίτερα κριτήρια και ρυθμίσεις για την πληρωμή αυτή. Επίσης, για το κατά πόσο θα πρέπει μόνο η ενεργή παραγωγή, πέμπτο ερώτημα. Εμείς δεν λέμε ότι οι μη δραστήριοι παραγωγοί θα πρέπει να παίρνουν τις πληρωμές ε, της ε, ΚΑΠ. Δεν είμαστε όμως πεπισμένοι ότι υπάρχει πρόβλημα στον ισχύοντα ορισμό των παραγωγών και ή της γεωργικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με, τον, ε, με το άρθρο 2 του κανονισμού. Ε, υπάρχουν παραγωγοί που ε, ιστορικά έχουν ε, δικαιώματα στην, ας πούμε που είχαν συγκεκριμένα, συγκεκριμένους αριθμούς ζώων με βάση τις, που είχαν υπολογιστεί στα αίτια αναφοράς και αυτά συνεχίζουν να πληρώνονται. Αυτό είναι μία όντως μία κατάκριση του, συστήμα, του συστήματος. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ε, οι πληρωμές να γίνονται με βάση την επιφάνεια. Εάν όμως ζητούν ε, πληρωμή και για επιφάνειες ε, όπου δεν ε, χρησιμοποιούνται για την γεωργία, τότε προφανώς δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε πληρωμή. Αν όμως παράγουν δημόσια αγαθά ή γεωργικά προϊόντα, τότε θα πρέπει να εισπράττουν τις, τα χρήματα ή επίσης όταν ακούμε ότι δίνονται χρήματα για γήπεδα του γκολφ ή τέλος πάντων για διαδρόμους αεροδρομίων ε, δεν καταλαβαίνω και το ξέρουμε αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί ε, τα κράτη-μέλη δεν ε, παρα, παρεμβαίνουν και δεν ορίζουν την, τη γεωργική γη. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν χρειάζονται νέοι ορισμοί ούτε για τους παραγωγούς ούτε για τη γεωργική χρήση. Εάν ε, πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, κυρίως αν αφορά το σύστημα άμεσων πληρωμών, είναι να γίνει ένα μεγαλύτερο πρασίνισμα. Και μια και ούτως ή άλλως ε, ε, εφόσον υπάρχει μια αποδέσμευση θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι ο παραγωγός μπορεί να παράγει προϊόντα ή περιβαλλοντικές υπηρεσίες δεν μπορούν να επιβάλλουμε να παράγουν και τα δύο. Ένα από τα δύο. Αρκεί. Πιστεύω ότι αν, αν θέλουμε να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο τον ορισμό, θα πρέπει ο παραγωγός να υποβάλει την αποδείξεις. Γι' αυτό θα εντείνει την γραφειοκρατία, θα είναι ένας εφιάλτης από τον οποίο δεν θα μπορούν να ξεφύγουν ούτε η παραγωγή ούτε οι δημόσιες υπηρεσίες. Ευχαριστώ τον καθηγητή κύριο Πίρτσιο Πύρολη. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντόουερ για 8 λεπτά. Thank you. Ευχαριστώ. Μιλώ για την ΑΡΚ σχετικά με τη, δηλαδή την ARC 2020 Agricultural and Rural Convention. Το ενδιαφέρον ε, είναι ε, να μπορέσει κανείς να ε, συνδυάσει και τις νέες χρήσεις των τροφίμων όπως τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και τα νέα τρόφιμα που απασχολούν ένα μεγάλο αριθμό ατόμων και ε, γι' αυτό στείλαμε ε, μία ανακοίνωση ε, γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά σε όλους τους ευρωβουλευτές και πρόκειται να την παρουσιάσουμε σε όλες τις γλώσσες σύντομα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει με τον πλανήτη και με τον κόσμο που ζει σε αυτόν και θα πρέπει πρέπει σύντομα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε εις ε, τις ε, προκλήσεις, να μειώσουμε ε, τα αέρια του θερμοκηπίου, να βελτιώσουμε τη βιοπικιλότητα, να σταματήσουμε την απώλεια βιοπικιλότητος, να έχουμε διατροφική ασφάλεια αλλά και ενεργειακή ασφάλεια σε έναν κόσμο με υπερπληθυσμό και να μειώσουμε τη φτώχεια και την την ανισότητα στην Ευρώπη και διεθνώς. Πιστεύουμε ότι για τα θέματα αυτά πρέπει να ρίξουμε ε, ένα νέο εξεταστικό μάτι εις ε, το συνολικό θέμα και ζητάμε να υπάρξει μία μετατόπιση εις ε, στα συστήματα τροφίμων και στην γεωργία συμμετέχοντας στη διαβούλευση που ξεκίνησε ο Επίτροπος Τσόλος ε, πριν από ένα χρόνο διαπιστώσαμε ότι ε, η ανακοίνωση αυτή και ε, το συνέδριο πέρυσι τον Ιούλιο έδειξε ότι υπήρξε μια μεγάλη ανταπόκριση εις το κοινό και χρειάζεται μια νέα κοινή γεωργική πολιτική η οποία να περιλαμβάνει υγιή και ασφαλή τρόφιμα και στήριξη ε, των αγροκτημάτων και ιδίως των μικρών γεωργών. Να προστατεύσουμε συγχρόνως το τοπίο και να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία. Η οργάνωσή μας ε, προσπαθεί να προωθήσει αυτό το θέμα και μέσω της ε, συμβάσεως ΑΡΚ προσπαθούμε να δώσουμε μία νέα νομιμοποίηση και στην γενική και γεωργική πολιτική και στον προϋπολογισμό της. Εξού και η γεωργία είναι το θέμα της πρώτης συνεδρίας, διότι πιστεύουμε ότι μέχρι το 2020 πρέπει να υπάρξει μία μετάβαση και σιγά σιγά να κινηθούμε από την ε, βιομηχανοποιημένη γεωργία στη βιώσιμη γεωργία παντού. Και αυτή η βιώσιμη γεωργία θα πρέπει ε, να βασίζεται στην αλληλεπίδραση των οικονομιών και ε, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανέφερε και ο κύριος Ντες, να χρησιμοποιεί τους πόρους, να σέβεται τη την ευημερία των ζώων, να μπορέσει να προωθεί την οικολογική ανανέωση και μεταρρύθμιση και ε, να μπορέσει να καταλήξει σε ε, νέες λύσεις περιβαλλοντολογικές και γεωργικές ε, για την Ήπεθρο και τις νέες περιοχές. Δηλαδή, με απλά λόγια πιστεύουμε ότι η στήριξη οικονομικά των γεωργών μέλλον μέλλον θα πρέπει να έχει σχέση με θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν θα επιτευχθούν μόνας τους από τις δυνάμεις της αγοράς. Χρειάζονται ενημερωμένα μέτρα της ρυθμίσεως της αγοράς. Είναι το δεύτερο θέμα που μας απασχολεί και θα πρέπει να δούμε Ποιο είναι το, ο, το ο, ο ποιο είναι το βασικό μας διακύδευμα, πώς πρέπει να αποδεσμεύσουμε τις άμασες πληρωμές, πώς θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τη χρήση του περιβάλλοντος, πώς θα στοιχηρίξουμε τις ε, μικρές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και πώς θα προωθήσουμε την ανάπτυξη, της, ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Για τις άμεσες πληρωμές προβλέπουμε μία συνέχιση των αμέσων πληρωμών βάσει σαφών προδιαγραφών βιωσιμότητος ή στην γεωργία χωρίς να υπάρχει αναφορά ή στις ιστορικές αποδόσεις με μια ισότητα πληρωμών μεταξύ των γεωργών των διαφόρων κρατών και ε, αντικατοπτρίζοντας την εθνική ε, αγοραστική δύναμη. Νομίζουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο. Θα πρέπει επίσης η ανώτατη πληρωμή ανά εκτάριο που θα αναφέρεται εις την πρώτη περιοχή ε, του, της κάθε εκμεταλλεύσεως και να μειώνονται όσο επεκτείνεται η ε, εκμετάλλευση αυτή. Με αυτό το σύστημα θα απαντήσουμε στο ερώτημα των μικρών γεωργών διότι θα πρημοδοτήσουμε αυτούς τους μικρούς γεωργούς αλλά θα πρέπει συγχρόνως να υπάρξει και ένας ορισμός τον οποίο υπενήχθηκε ο κύριος Ντες δηλαδή τι εννοούμε όταν μιλάμε για μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ένα, με, ε, ένα σύνολο μέτρων υπό τον δεύτερο πυλό θα μπορέσει να βοηθήσει τους μικρούς γεωργούς σε λιγότερο προνομούχες περιοχές, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για να υπάρξει μία διαδοχή στι ε, τα, στο, ε, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να μπορέσουν να έχουμε σωστή σήμανση των γεωργικών προϊόντων και όσον αφορά τους ενεργούς γεωργούς πιστεύουμε ότι όλοι είτε εργάζονται ε, πλήρως είτε με, με μερική απασχόληση θα πρέπει να έχουν ε, πρόσβαση στις άμεσες πληρωμές διότι έτσι θα υπάρξει ε, τη, η δυνατότητα να έχουμε τη δυνατότητα για όλους να είναι εκλέξιμοι από περιβαλλοντολογική πτυχή και εκτός εάν ε, ε, αυτό δεν θα συμπεριλαμβάνει τους γεωκτήμονες εκτός αν ο κύριος Πέσιο Παρόλη ε, υπενήχθηκε ότι και οι γεωκτήμονες εργάζονται στις εγκαταστάσεις τους. Με συγχωρείτε πρέπει να κλείνετε λέγει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Ντόουερ. Θα πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο γιατί αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σπάν, ο οποίος εκπροσωπεί το, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των ε, συνδικάτων, των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Επίσης θα ήθελα να χαιρετήσω και την παρουσία των Ιταλών ε, που βρίσκονται στην αίθουσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ότι δεν εκπροσωπούνται ε, εδώ μόνο ε, τα Ιταλικά συνδικάτα αλλά ε, όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ευρώπης και από το Βορρά και από τον Νότο διότι δείχνει ότι η συζήτησή μας έχει ένα μέλλον. Έχουμε πάνω από 7 εκατομμύρια εργαζομένους στο γεωργικό τομέα της Ευρώπης. Πληττόμεθα από τις αποφάσεις και γι' αυτό περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την εισήγηση του κυρίου Ντες ο οποίος θα μπορέσει να μας παρουσιάσει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές αλλά εδώ αυτό το θέμα δεν είναι σημαντικό μόνο για τους εργαζομένους ή την Ήπεθρο αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε σε αυτή τη νέα Ευρώπη διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει μεγάλο ρόλο εις ε, τις χώρες κατόπιν της διευρύνσεως και πρέπει να διέπει την όλη διαδικασία δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν να δω, δούμε όλοι πώς τοποθετούμεθα σε αυτή τη νέα Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δούμε αν θεωρούμε ότι οι κανόνες ε, του οικοδομήματος αυτού είναι σωστοί. Και ο ίδιος ο κύριος ε, Ντες ανέφερε ότι σε ορισμένες χώρες υπάρχει μία σημαντική μείωση του ενδιαφέροντος και της στήριξης του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και ιδιαίτερο στον τομέα της γεωργικής πολιτικής. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν δεν εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες της γεωργικής πολιτικής στα νέα κράτη ε, θα υπάρξει μία έξαρση του εθνικισμού ε, και γι' αυτό το λόγο και μόνο θα χρειαζόταν ε, ένα σαφής κανόνας για την ε, ε, σωστή και τακτική μεταφορά των κανόνων αυτών και της νομοθεσίας ε, ε, στα νέα κράτη όπως άλλωστε υπάρχει και τώρα μεταξύ ε, βορείων κρατών και της Ελλάδος παραδείγματος χάρη πρέπει λοιπόν ο καθένας να γνωρίζει που βρίσκεται η θέση του στο μελλοντικό οικοδόμημα της γεωργίας της Ευρώπης και αυτό είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο όσους ασχολούνται με τη γεωργία αλλά με όλους που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κοινοβούλιο και ε, ήδη ακούσαμε διάφορα σχόλια από αυτού. Όπως σας είπα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ε, ε, θέσεων εργασίας που κατεστράφησαν στις νέες χώρες. Η Ουγγαρία είχε θαυμάσια σαλαμοποίια. Όλοι ήταν, τα ουγγρικά σαλάμια ήταν γνωστά αλλά τώρα έχει καταστραφεί η παραγωγή αυτή και δεν είναι δυνατόν επιπλέον να κρατήσει κανείς κανείς τις εκτάσεις που είχε στο γεωργικό τρομέα και γι' αυτό και μίλησα για μία νέα μέθοδο. Με την πολλαπλή συμμόρφωση επίσης χάθηκαν πολλές θέσεις εργασίας και ε, γι' αυτό ε, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι με τις άμεσες πληρωμές 20% των επιχειρήσεων παίρνουν τον 80% των πληρωμών παρόλο που είναι μία, ένα αποτέλεσμα της απελευθερώσεως η οποία υπήρξε. Ε, ίσως δεν έχω ακόμη σχολιάσει τα, τις έξι ερωτήσεις που έθεσε ο εισηγητής αλλά ήθελα να σας πω ότι και στον οικολογικό τομέα θα πρέπει να υπάρξει προσαρμοστικότητα και γι' αυτό χρειάζεται και ανάπτυξη της εκπαιδεύσεως εξού και πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι στον ε, γεωργικό χώρο άντρες και γυναίκες πρέπει να έχουν πρόσβαση εις ε, την ε, συγκεκριμένη εκπαίδευση. Όσον αφορά την, πρόσταση, την οδηγία της προστασίας της εργασίας δεν βλέπουμε να έχει μετατεθεί στη γεωργία που είναι ένας πολύ επικίνδυνος και παρόλο που υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες μέσω της cross compliance βλέπουμε ότι εδώ ο κάποιος μπορεί να πει ότι όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ περίπλοκα και υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία και ε, αν κάποιος ε, έχει ως μεγάλο εισόδημα δημόσιες ε, εισφορές ε, τότε ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα μειωθεί και για αυτούς που εξαρτώνται από, ε, από τη γραφειοκρατία μία μείωση του γραφειοκρατικού φορτίου ε, πρέπει να δούμε ε, λοιπόν ότι δεν πρέπει μόνο να προστατεύσουμε παραδείγματο χάνει τις αγελάδες αλλά να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό το χώρο. Είναι 15% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, και δεν μιλάμε μόνο για τους απασχολούμενους αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει υπάρξουν συζητήσεις για το πώς θα προσαρμοστούμε, μέτρα για, το, για να προσαρμοστούμε, διότι είδαμε ότι σε διάφορες χώρες τα νέα μέτρα είχαν δραματικές επιπτώσεις. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει για την προστασία του εδάφους και του ύδατος και όντως πρέπει η νέα γεωργική πολιτική να μας μας βοηθήσει να στηρίξουμε και να προστατεύσουμε καλύτερα το περιβάλλον για τα υπόγεια ύδατα και για την διατήρηση υγιών εδαφών. Ε, είμαστε ε, κατά ε, ενός συνδυασμού διότι το ερώτημά μας είναι να γνωρίζουμε πώς πρέπει να εργαστούμε και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι ε, κοινωνικά ασφαλισμένοι και κατά μέσον όρον θα πρέπει ε, να υπάρξει μία κάλυψη ε, μέσω άλλων δυνάμεων παραδείγματο χάρη των επιχειρήσεων διότι βλέπω ότι τώρα αυτό είναι 50%. Έχω στοιχεία τα οποία θα δώσω γραπτός διότι ε, πρέπει να περιορίσω το χρόνο ομιλία μου. Ε, Γενικώ όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι μέλος της προτάσεως που διαμορφώνουμε και γι' αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι πληρωμές Επίση, Επίσης οι γεωργοί είναι άτομα που έχουν επιμορφωθεί στο τομέα τους και θα πρέπει ε, να γνωρίζουν επίσης τους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής και ε, η οικογένεια των γεωργών δεν πρέπει να ξεχαστεί στα μελλοντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σπάνα. Ο τελευταίος ομιλητής, η κυρία Μένα Φρίδεν της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα ε, τροφίμων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το πρώτο πράγμα νομίζω που πρέπει να αναφέρω είναι ότι η γεωργία είναι εξαιρετικά σημαντική για την βιομηχανία μου, τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών χρησιμοποιούμε το 70% αυτών που καλλιεργεί η Ευρωπαϊκή Γεωργική Κοινότητα. Έξω και παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά και από πολύ κοντά αυτά που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της ε, γεωργικής πολιτικής. Ε, η γεωργία παρέχει λοιπόν πρώτες ύλε στην αλυσίδα τροφίμων και είναι πάρα πολύ σημαντική η γεωργοδιατροφική βιομηχανία είναι μεγαλύτερη στην Ευρώπη, ψηλά ποσοστά απασχόλησης, μεγάλη προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή οικονομία υπό οικονομικού όρου, η Ευρωπαϊκή Γεωργία και η βιομηχανία των τροφίμων είναι πάρα πολύ σημαντικοί τομεί που παρέχουν απασχόληση σε 17 εκατομμύρια ανθρώπου ε, και στα 27 κράτη-μέλη βέβαια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μακροχρόνια βιωσιμότητα των δύο λοιπόν αυτών κλάδων ε, συμβαδίζει, πηγαίνει χέρι με χέρι. Και νομίζω ότι η προσέγγιση που τουλάχιστον εμεί θα θέλαμε να δούμε από την βιομηχανία τροφίμων είναι αλυσιδωτή προσέγγιση αν θέλετε. Δηλαδή να μην εξετάζεται από ξεχωριστή σκοπιά η γεωργία αλλά θα πρέπει να δοθεί συνολικά στο πλαίσιο της όλης αλυσίδας από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή δηλαδή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε την ασφάλεια των τροφίμων ως μείζωνα πρόκληση. Και έχει βέβαια ε, καταστεί και ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Και βέβαια αυτό συμβαδίζει και με την αηφορία, τη βιωσιμότητα. Συμβαδίζει επίσης με την πρόληψη των υπερβολικών διακυμάνσεων των τιμών, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Και βέβαια η ανταγωνιστικότητα του κλάδου είναι πολύ σημαντική. Και βέβαια η πρόθεση της έρευνας και της καινοτομίας, γιατί η ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι κάτι που μπορεί να το δούμε απομονωμένο αλλά ε, στο πλαίσιο όλων αυτών των άλλων ζητημάτων, βιωσιμότητα, διακυβάσεις τιμών, ανταγωνιστικότητα, έρευνα, καινοτομία. Και αν τα πετύχουμε όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό θα αποβεί προς όφελος όλη τη τροφική αλυσίδα και όλης τη αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτή είναι η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί για την ε, αλυσίδα εφοδιασμού. Νομίζουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιες ε, σημαντικέ αρχές. Στη δική μας νομοσπονδία δεν εξετάζουμε με λεπτομέρειες, ούτε μπορούμε να ορίσουμε τι θα πει ενεργός αγρότης, πώς ορίζεται. Αυτές τις λεπτομέρειες αφήνουμε στους συναδέλφους μας από την κόπα ΚΟΣΕΓ. Η CIAA, όπως γνωρίζετε, η δική μας νομοσπονδία, απαρτίζεται και από πολύ μεγάλες αλλά και από μικρές επιχειρήσεις, εθνικές ομοσπονδίες τροφίμων και ποτών, από όλες τις χώρες και από διάφορους τομείς, γαλακτοκομικό, ζάχαρη και όλους τους άλλους τέλος πάντων. Επομένως, δεν είναι πολύ εύκολο να κάνουμε αυτές τις πολύ ενδελεχείς συζητήσεις. Εκπροσωπούμε βορρά, νότο, μικρές, μεγάλες επιχειρήσεις, παραγωγή, μεταπίση. Όπως καταλαβαίνετε αγωνιζόμαστε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για όλες αυτές τις πάρα πολύ αναλυτικές συζητήσεις. Αυτό που μπορούμε πάντως να πούμε και συμφωνούμε όλοι από αυτού είναι ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να εγγυάται τον ισότιμο ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εναρμόνιση λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προωθεί να ενισχύει την παραγωγή εντός ευρωπαϊκής ένωσης ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και να ε, ανταποκριθούμε στις προκλήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει να υπάρχουν εργαλεία για την καταπολέμηση όπως είπα των πολύ σημαντικών διακυμάνσεων των τιμών που επηρεάζουν πολύ αρνητικά και θεωρούμε βέβαια ότι αυτό θα πρέπει να σχετιστεί και με τον αγοροκεντρισμό Πιστεύουμε ότι η περαιτέρω πρόθεση και υποστήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των βιώσιμων και αποδοτικών για τους πόρους πρακτικών είναι θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη αλλά θα πρέπει να λέμε υπόψη τις περιβαλλοντικές και άλλες προκλήσεις. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι ο γεωρικός περιπολισμός φυσικά και θα πρέπει να δίνει τα μέσα στην κοινή γεωρική πολιτική ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους που έχουν τεθεί. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα δύο ερωτήματα, μάλλον τα πολλά ερωτήματα του πρώτου τμήματος για τις άμεσες πληρωμές. Για μας έχουν να παίξουν ρόλο και οι δύο πυλώνες, και ο πρώτος και ο δεύτερος, για τη βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Η βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής περιλαμβάνει την οικονομική βιωσιμότητα, την κοινωνική ευθύνη και την ε, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και όλα τα μέτρα θα πρέπει να φροντίσουν να εξασφαλίσουν ένταση προβλεψιμότητας για τους αγρότες. Θα πρέπει να έχουν ένα μακρόπνο όραμα για μια μακροπρόθεσμη συμπεριφορά και θα πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ελκυστικού επιχειρηματικού κλίματος. Το ανέφεραν και κάποιοι άλλοι ομιλητέ. Πράγματι, η πολιτική για την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να προσελκύσει του νέου αγρότε και να αναστρέψει την σημερινή τάση όπου πάνω από 50% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν ε, διευθυντές ηλικίας άνω των 55 ετών. Πρέπει να ε, εμφυσίσουμε νέα πνοή, δίνοντας, μεταγγίζοντας, αν θέλετε, νέο αίμα στη γεωργία. Τώρα, οι άμεσες πληρωμές είναι πάρα πολύ ε, συναρπαστικό θέμα που θέλω να πω ότι είχαμε και μια συζήτηση πάρα πολύ ζωντανή ενδιαφέρουσα στην Συνομοσπονδία μας και νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε εν είναι βιώσιμη ε, προμήθεια, αλλά κατά περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Η εφαρμογή των βιώσιμων για το περιβάλλον πρακτικών και αποδοτικών πρακτικών είναι στον πυρήνα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη μακροπρόθεσμα αν δεν δοθεί έμφαση περισσότερη στι βιώσιμε γεωργικέ πρακτικέ. Και εδώ αναφέρομαι στην την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων συγκεκριμένα, κλιματική αλλαγή, βιοπικιλότητα. Για να μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε όλα αυτά, παραλαμβάνω, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης τροφικής αλυσίδας, Ξέρετε ότι ενώσαμε τις δυνάμεις μας και με τους άλλους παράγοντες της ε, τροφικής αλυσίδας και έχουμε δημιουργήσει και το ε, γύρο τραπέζης για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση είναι πολύ επιτυχή η όλη μα προσπάθεια προ επίτευξη των στόχων μα. Με τα χαρά το λέω Με τα χαρά στο λέω αυτό. Θα σταματήσω εδώ. Ελπίζω να απάντησε σε κάποιε από τι ερωτήσει σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, όλους σας. Ε, σεβαστήκαμε απόλυτα το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μα. Τώρα ε, ξεκινάει ο διάλογος με τα μέλη της Επιτροπής. 11 συνάδελφοι από διάφορες πολιτικές ομάδες έχουν ζητήσει το λόγο. Σας ζητώ το, να σεβαστείτε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, δύο λεπτά ο καθένας, για να μπορείτε και εσείς ε, να θέσετε την ερώτησή σας και τα μέλη του πάνελ να απαντήσουν. Και θα ήθελα να διευκρινίσετε σε ποιον ομιλητή κάνετε την ερώτηση, εάν και εφόσον απευθύνεστε κάποιο συγκεκριμένα. Ο κύριος Πίτερ Γιάρ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ερωτήσεις μου απευθύνονται σε όλους τους ομιλητές. Και εδώ πρόκειται για τις άμεσες πληρωμές και την ε, γενική αιτιολόγηση για τις άμεσες πληρωμές που στην αρχή ήταν η πολλαπλή συμμόρφωση. Ε, το ερώτημα είναι πρέπει να παραμείνουμε στο ίδιο σκεπτικό ή χρειαζόμαστε και άλλες αιτιολογίες για τις άμεσες πληρωμές διότι ε, επίσης άλλη ερώτηση πιστεύετε ότι δικαιολογείται το ύψος των αμέσων πληρωμών πρέπει να αυξηθεί, να μειωθεί ή να εκεί. Ε, τρίτον, ποια είναι, ποιος είναι ο ιστορικός συσχετισμός και πώς επιδρά. Ε, τέταρτον, επειδή ε, όλοι κάπως ε, ε, δεν ήταν σαφείς στην ερώτηση αυτή πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει μία αιτιολογημένη κατανομή ανακράτος και πέμπτον ποια άμεσης πληρωμές θεωρείτε ότι είναι αιτιολογημένες εντός μίας, μίας χώρας μέλους. Ε, μετά, ε, όσον αφορά το ανώτατο όριο, για αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι είναι δικαιολογημένο να υπάρχει ένα πλαφόν, ένα ανώτατο όριο, ε, έχετε κάποια οικονομική ή λογική αιτιολογία για να καθορίσετε το πλαφόν. Γιατί δηλαδή πρέπει να είναι 50.000 ευρώ ή 150.000 ευρώ. Υπάρχει μία λογική αιτιολογία και θα θέλατε η κάλυψη αυτή να συνδυαστεί και με άλλα κριτήρια και τέλος πιστεύετε ότι η σχέση μεταξύ ε, πρώτου και δευτέρου πληρώνα πρέπει να αλλάξει πρέπει ε, να ε, αυξηθεί να μειωθεί η συμμετοχή του πρώτου πυλώνα σε σχέση με το δεύτερο πυλώνα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ομιλητές για όλα όσα είπαν, αλλά και να εκφράσω και την απογοήτευσή μου, διότι θέσαμε πέντε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις και εγώ περίμενα πέντε συγκεκριμένες αντικειμενικές απαντήσεις. Και με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν νομίζω ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Θέλαμε να ξέρουμε αν συμφωνούσαν ή όχι με, την, με τις άμεσες πληρωμές. Οι περισσότεροι είπαν ναι και μετά μας είπαν για την ισότιμη κατανομή τι λέτε. Άλλοι είπαν ναι, άλλοι είπαν όχι. Για, την, για το πρασίνισμα, ε, εντάξει υπάρχει μια γενικευμένη συμφωνία ίσως να υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει ανατοτόριο για τις, ε, για τις πληρωμές, αλλά για το τελευταίο ερώτημα δεν είχαμε καμία σαφή απάντηση. Να κάνω μία άμεση ερώτηση, εγώ και συγκεκριμένη. Στην επόμενη μεταρρύθμιση το θέμα των άμεσων πληρωμών είναι κέριο ερώτημα. Επομένως, αν όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν άμεσες ε, πληρωμές σε όλους τους παραγωγούς, ήθελα να ξέρω εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η βάση για τον υπολογισμό αυτών των άμεσων πληρωμών. Θα πρέπει να ισχύουν περιβαλλοντικά κριτήρια, θα πρέπει να υπάρχουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή δημιουργία θέσεων απασχόληση ή κάτι άλλο. Ευχαριστώ Λουίσα. Ο Αντιπρόεδρος Ζωζέ Μπουβέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ε, στην ερώτηση που θα θέσω θέλω να απευθυνθώ εις ε, την ε, διατροφική βιομηχανία και θα ήθελα να ξέρω αν στα πλαίσια αυτής της πολιτικής σκοπεύετε να λάβετε μέτρα κατά τρόπον ώστε ε, να μην ε, πληρώνονται ποτέ οι γεωργοί κάτω από το κόστος παραγωγής τους διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει παραγωγή ε, εάν η διατροφική βιομηχανία η βιομηχανία τροφίμων και τα, οι μεγάλες αλυσίδες δεν καλύπτουν τουλάχιστον τα έξοδα παραγωγής των γεωργών. Μετά, το δεύτερο μου ερώτημα αναφέρεται στους μικρούς γεωργού και αναφέρομαι και στην Κοπά και στην κυρία Καπεσίνα και θα ήθελα να πω ότι γνωρίζετε ότι σήμερα εάν να πάρουμε ένα ορισμό βάσει της επιφανείας 5 εκταρίων το, η με κάτω από 5 ε, εκτάρια είναι 12,5 εκατομμύρια στην ε, Ευρώπη. Υπάρχει το θέμα όμως της επιφανίας ε, του τζίρου και των ενισχύσεων. Πώς λοιπόν θα στηρίξετε και θα ενισχύσετε στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής τα 12,5 εκατομμύρια άτομα αυτά. Επίσης η νομιμοποίηση της ε, γεωργικής πολιτικής. Αυτό είναι, ε, τι, είναι έτοιμος να καλύψει ο πολίτης ε, για το κόστος αυτό. Εάν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων που ενισχύονται και άλλες που δεν ενισχύονται, πώς θα προχωρήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσει. Ευχαριστώ Ζωζέ. Και τώρα ο κύριος Λόσεβιτς. Βλάσεκ Λόσεβιτς. Και εμένα το ερώτημά μου αναφέρεται στις άμεσες πληρωμές διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένως έχει ε, αναφερθεί σε μια πιο δίκαια κατανομή των αμέσων πληρωμών και είναι προφανές ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να διατηρηθεί και όπως πολλοί ομιλητές είπαν είναι δύο αντικρουόμενα συστήματα. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα συστήματα αυτά, αυτό ρωτούμε όλοι, διότι αν υποθέσουμε ότι υπάρξει ε, μια κοινή γεωργική πολιτική για τα επόμενα έτη πώς θα κατανείμουμε τη χρηματοδότηση για να αποφύγουμε τριβές σε ορισμένα κράτη-μέλη. Επίσης ε, θέλω να κάνω και την ε, ακόλουθη ερώτηση. Πώς προβλέπετε να λυθεί αυτό το πρόβλημα και αν μπορώ θα ήθελα να προτείνω ε, μία πιο συγκεκριμένη απάντηση διότι όλοι οι γεωργοί θα έπρεπε να την χάνουν μια αντικειμενική αντιμετωπίσεως. Ε, τι πιστεύετε για αυτή την πρόταση ή πιστεύετε ότι αν πρέπει να υπάρχουν ίσες άμεσες πληρωμές σε όλη την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση θα συμφωνήσετε. Ευχαριστώ. Ο Άλφρεντ Ρούμπιν έχει το λόγο τώρα. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγεται σαφέστατα ότι το σύστημα των άμεσων πληρωμών πρέπει να αναθεωρηθεί και το σύστημα αυτό πρέπει να συνδέεται σε με ένα νέο σύστημα, δηλαδή μια, μια νέα κατανομή με βάση τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Θα πρέπει επομένως αυτό το σύστημα να στηρίζεται σε, οικονομικούς, σε οικονομικά κριτήρια και σε περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτό το σύστημα πρέπει να είναι ευανάγνωστο αν θέλετε και για τους παραγωγούς αλλά και για τους φορολογούμενους. Όλα αυτά μένα με βρίσκουν σύμφωνο. Το πρόγραμμα, το μελλοντικό πρόγραμμα της Κομισιόν το 2013 προβλέπει τρία σενάρια για την χρησιμοποίηση των δύο πυλώνων. Συμφωνώ απόλυτα με το γεγονός ότι στο μέλλον χρειαζόμαστε δύο πυλώνες. Στην χώρα μου, ε, εγώ είμαι από τη Λιθουανία, στη Λετωνία, συγγνώμη, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τους δύο πυλώνες. Όμως για μας, για τη Λετωνία, αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει η αναθεώρηση των, ε, για τις άμεσες πληρωμές. Η Λετωνία προτείνει το εξής. Στο μέλλον, οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν δύο τμήματα το ένα τμήμα θα πρέπει να αφορά τα μέσα και οι ενισχύσεις για την διατήρηση των γεωργικών γεών και το δεύτερο τμήμα θα πρέπει να είναι η βοήθεια, η ενίσχυση της γεωργίας. Και εδώ ισχύουν ε, ας πούμε κριτήρια όπως το ΑΕΠ ε, ή να χρησιμοποιούμε και ένα συντελεστή για να δούμε κατά πόσον τα μέσα τα οποία δίδουμε ε, είναι επαρκή ή όχι. Μετά θα πρέπει να γίνουν βέβαια και κάποιες προσαρμογές για να γίνει μια προσάυξη των ε, ενισχύσεων. Επίσης ε, πρέπει να διατηρηθούν οι ενισχύσεις για τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές μετά το 2012 ο κύριος Τζοβάνι Λαβία. Εδώ είμαστε μπροστά σε μία ανευθυνότητα μέσα από τους κανόνες που θα διέπουν την μελλοντική ΚΑΠΑ ζητάμε από τον κύριο Κόλτερ να μας δώσει κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις που θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε την έκθεση που θα συντάξουμε το σημερινό σύστημα για την χορήγηση των πληρωμών, άμεσο πληρωμών, στηρίζεται σε ένα ιστορικό ε, κριτήριο των πληρωμών. Ε, μας είπανε όμως ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη καθυστέρηση. Χρειάζεται όμως για να περάσουμε σε ένα νέο σύστημα να έχουμε και μια μεταβατική περίοδο. Πόσο μεγάλη, πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η μεταβατική περίοδος για να μην πληγούν οι παραγωγοί. Επίσης, η γεωργική η γεωργία της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις και όσον αφορά το μέγεθος και όσον αφορά την παραγωγή κτλ. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την, τις γεωργικές επιφάνειες. Κάποιος μας, ο εισηγητής μας είπε ότι 10 εκτόρια, 10 εκτάρια μπορεί να είναι μια μικρή γεωργική εκμετάλλευση. Όμως μπορεί ε, αν έχουμε μια εντατική παραγωγή να θεωρηθεί και μεγάλη η εκμετάλλευση. Επομένως, στα διάφορα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, έχουμε και συμπληρωματικά κριτήρια. Ας πούμε η παραγωγή, ε, η εργασία που έχει επενδυθεί, η αξία της απόκτησης της γης στις διάφορες ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαν αυτά να αποτελέσουν συμπληρωματικά κριτήρια για την χορήγηση των άμεσων πληρωμών στα κρατημέλη και στο εσωτερικό των κρατών, μελών. Ο κύριος Σικυριέσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Το ε, έργο και η ζωή του ανθρώπου συνδέεται με τη βιολογία και τα ζώντα ζώα. Άρα τον τομέα αυτό δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ας δούμε τι έχει επιτύχει μέχρι στιγμής η κοινή γεωργική πολιτική. Σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα οι αγρότες ό,τι αφορά την ηλικία, το εισόδημα, η νεολαία, τι κάνει. Όλες ε, τις πληροφορίες της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι αγρότες ε, πώς τις αντιλαμβάνονται και τι κοστίζει τελικά η κοινή αυτή πολιτική. Και τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Παντού υποστηρίζεται η ανάπτυξη της γεωργίας. Δείτε τον ΠΟΕ. Η γεωργία εκεί μάλλον φαίνεται να είναι στο στρατόπεδο των ιτημένων. Η... Είχαμε την ΚΑΠ το 2002, ε, ε, πρώτο στάδιο, 2003 μεταρρύθμιση νέοι όροι και αυτό χωρίς να ληφθεί υπόψη διεύρυνση. Οι χώρες της διεύρυνσης δεν ωφελήθηκαν. Μιλάμε λοιπόν για μια δωδεκαετία, με χρονική περίοδο για τη Γεωργία. Έχουμε πάντως κοινή γεωργική πολιτική. Έχουμε νέα αγορά, Έχουμε κοινωνικά πρότυπα, περιβαλλοντικά, ποιοτικά πρότυπα και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι υφίστανται, υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Όμως οι αγρότες μπορεί να ζουν στην Πολωνία για παράδειγμα, αλλά αγοράζουν τα λοιπάσματά τους στη Γερμανία. Και δεν νομίζω ότι χωρεί αμφιβολίας ότι και στην διαδικασία της διεύρυνσης έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις. Ας δούμε τώρα τι σημαίνει με τους μικρούς αγρότες. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις απασχολούν λίγα άτομα. Φαίνεται ότι ίσω να μην απαιτήσουν ε, στήριξης. Δυστυχώ έκλεισε το μικρόφωνο. Η Εράνθα Γκαρθία. Ευχαριστώ πολύ. Έχω να δώσω και εγώ κάποιες ε, ιδέες. Σίγουρα η αναδιανομή των ενισχύσεων τη κοινή γεωργική Πολιτική είναι αναπόφευκτη. Αλλά δεν θα πρέπει αυτό να οδηγήσει σε τραυματικέ καταστάσει που θα θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα εφιστάμενων εκμεταλλεύσεων. Να μην χάσουμε τις ήδη φυστάμενες αφού ούτε καν ανακυκλώνονται οι επιχειρήσεις. Τώρα τα συστήματα παραγωγής, ειδικά συστήματα παραγωγής, πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά δεν άκουσα ούτε μία κουβέντα γι' αυτό. Υπάρχουν ε, κάποιες, ε, ε, υπάρχει εντατική γεωργία η οποία όμως πληρεί τις προϋποθέσεις αλλά αν δεν λάβει ενισχύσεις θα εξαφανιστεί. Επίσης ό,τι αφορά το modulation, αυτή τη διαβάθμιση, εγώ νομίζω πρέπει να εξαλειφθεί από την ορολογία, τη φρασιολογία της κοινή γεωργικής πολιτικής γιατί μπορεί να προκαλέσει μεγάλες εντάσεις και κατά την ανακατανομή των ενισχυών και ουσιαστικά συνιστά μια κρυφή αν επανακρατικοποίηση. Θέλω να ακούσω τι έχετε να πείτε από αυτόν. Τώρα σε ό,τι αφορά τα, πλα, τα πλαφόν θα πρέπει να βασιστούν ε, σε συγκεκριμένους όρους και θα πρέπει να βάλουμε λέξεις, όρους, ετικέτες. Απασχόληση που παράγει, που γεννά κάθε εκμετάλλευση κτλ. Και θα ήθελα επίσης να μας πείτε και κάποια πράγματα για τη διοικητική απλούστευση. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει οι αγρότες να τρομάξουν μπροστά ε, στον όγκο της γραφειοκρατίας που συνιστά η κοινή γεωργική πολιτική για αυτούς. Ξέρουμε ποιες είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα άμεσε πληρωμέ πρώτο πυλώνα συνολικά νομίζουμε ότι πρέπει να χρηματοδοτούνται 100% από τον κοινοτικό προπολογισμό. στον πρώτο πυλώνα επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα προς όλους τους εμπειρογνώμονες. Γιατί Όλοι αναφέρατε κάποια αντικειμενικά τελικά κριτήρια για να ορίσετε τις άμεσες πληρωμές. Μετά από διαβουλεύσεις με τους αγρότες γίνεται πρόταση για τον καθορισμό διαφόρων, περισσότερο του ενός αντικειμενικών κριτήριων. Πρώτον, η έκταση που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, ΑΕΠΑ, ανακάτοικο κατά κεφαλήν και τρίτον, κόστος συντήρησης των γεών συμπαρελαμβανομένης εκμετάλλευση της τεχνικής καυσίμων εργατικού δυναμικού της γεωργικής εκμετάλλευσης. Θεωρείτε ότι πρόκειται για σημαντικά κριτήρια για την επιτεύξη των ε, στόχων, των στόχων για πιο ακριβοδίκαια εισοδήματα και για πιο ακριβοδίκαια υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει ένα κατώτατο όριο εγγυημένο με βάση τα μέσα επίπεδα στήριξης. 75% τουλάχιστον εκτιμούν οι αγρότες. Εσείς θεωρείτε ότι είναι δίκαιη η πρόταση αυτή. Επίσης θα πρέπει να ορίσουμε το πλαφόν Δηλαδή τη στήριξη ανά εκτάριο, τη βοήθεια, την ενίσχυση ανά εκτάριο στο τάδε ήδη ένα κράτος μέλος. Κατά την άποψή σας, αντιστοιχεί, ε, συνάδει με τη μελλοντική κάπα αυτή η πρόταση και τέλος, ό,τι αφορά τη μεταβατική περίοδο. Όπως γνωρίζετε, τα νέα κράτη-μέλη ήδη από το 2004 και μετά ζουν μέσα σε μια μεταβατική περίοδο. Το 2013 έχουμε κάποιους υπολογισμούς που θα ισχύουν 100% για όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τα ιστορικά στοιχεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο σημεία. Το πρώτο σημείο αφορά στη δίκαιη κατανομή των πόρων. Η ίδια η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η δίκαιη κατανομή δεν σημαίνει ίση κατανομή των ενισχύσεων και ότι η ενιαία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στρεματική ενίσχυση, flat rate, δεν συνιστά λύση. Είναι βεβαίως γνωστές οι ουσιώδεις διαφορές που υφίστανται μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, και κρατών μελών ως προς το κόστος παραγωγής, τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη συμβολή της γεωργίας στην απασχόληση και στην οικονομία ποια κριτήρια πρέπει να προκριθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις σωσάνω διαφορές. Σημείο δεύτερον, η Κομισιόν εισηγείται τη μεταφορά ορισμένων μέτρων από το δεύτερο στον πρώτο πυλώνα, όπως αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, μέτρα για μηνυκτικές περιοχές. Θεωρείται ότι θα πρέπει η μεταφορά αυτή να συνοδευτεί από την αντίστοιχη ανακατανομή πόρων redistribution από τον δεύτερο προς τον πρώτο πυλώνα. Οι ερωτήσει μου ε, απευθύνονται σε όλους τους εκπροσώπους των αντιπροσωπευτικών ε, φορέων, στους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία τους και για τις εισηγήσεις τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ George. Ο τελευταίος από τους 11 η τελευταία μάλλον η Διάννα, Διάννα Τόντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ομιλητές Καταρχήν αναφέρομαι στην πρώτη ερώτηση που έχουμε στον κατάλογο, δηλαδή πώς οι πληρωμές του πρώτου πυλώνα μπορούν να κατανεμηθούν πιο δίκαια. Ε, είναι κρίμα που δεν είχαμε περισσότερους ορισμούς για να διευκολύνουμε τους φιλοξενούμενους μας και εγώ δεν νομίζω ότι σε αυτή την Επιτροπή υπάρχει διαφάνεια και σαφήνεια, οπότε ε, θα πρέπει να δώσετε το παράδειγμα στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μία διευκρίνηση. Θα ήθελα να ξέρω ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια για αυτές τις άμεσες πληρωμές ε, και αν πρέπει να περιλάβουμε μία μεγάλη μεταβατική περίοδο περίοδο αν πρέπει να λάβουμε υπόψη την αξία των εκτάσεων και ούτω καθεξής. Δηλαδή αμφισβητώ πολύ την πορεία την οποία διαγράφουμε αυτή τη στιγμή. Ε, όσον αφορά την πιο περιβαλλοντολογική αντιμετώπιση των πληρωμών από τον πρώτο πληρών, μήπως έτσι θα είμαστε πιο εκτεθειμένοι στην πολλαπλή συμμόρφωση που είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και θα ήθελα να το σχολιάσετε διότι εμείς δεν θέλουμε ε, να έχουμε και περιβαλλοντολογική γραφειοκτατία εκτός από τη γεωργική. Όσον αφορά την νομιμοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής, θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας. Θεωρώ ότι είναι μία νόμιμη πολιτική. Δεν χρειάζεται να γίνει η κοινή γεωργική πολιτική ούτε κοινωνική ούτε οικονομική. Χρειάζεται για να παράγουμε στην Ευρώπη τρόφιμα και να εξυπηρετούμε τον καταναλωτή. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς εσείς αντιμετωπίζετε και αυτή την νομιμότητα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχουμε δύο λεπτά για όλα τα μέλη του πάνελ για να απαντήσουν. Και μετά περνάμε στο δεύτερο γύρο που θα έχετε πάλι χρόνο για να μιλήσετε. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον πρόεδρο της ΚΟΠΑ, τον κύριο Walsh. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, προφανώς δεν μπορώ να απαντήσω ε, σε όλες τις ερωτήσεις αυτές για δύο λεπτά. Ε, θα ήθελα όμως να, πω, να ευχαριστήσω την κυρία Ντότζ ε, γιατί είπε αυτό το οποίο ήθελε να πω και εγώ. Αν, είχαμε, ήταν εύκολο να είχαμε αντικειμενικά κριτήρια θα τα είχαμε βρει μέχρι τώρα. Αυτό θέλουμε όμως. η γεωργία, αυτό το οποίο θέλουν οι παραγωγοί, αυτό το οποίο θέλουν είναι να κερδίσουν το εισόδημά τους από την αγορά, από την πώληση δηλαδή των προϊόντων που παράγουν. Και αυτό κάναμε ε, μέχρι ότου άλλαξε η ΚΑΠ στις αρχές του 90, όπου εισήχθη αυτό το σύστημα ε, των άμεσων πληρωμών, το οποίο συνδυόταν με την παραγωγή καταρχάς. Και μετά, όπως ξέρουμε, άλλαξε το σύστημα και είχαμε ένα σύστημα το οποίο συνδυόταν με την ιστορική παραγωγή. Και εδώ ε, έχουμε την άλλη, άλλη μεταρρύθμιση και η πρώτη ερώτηση ήταν ποια θα ήταν, ποια θα μπορούσαν να είναι τα νέα κριτήρια για να δικαιολογήσουν τις πληρωμές θα κόστιζε πολύ λιγότερο στον Ευρωπαίο φορολογούμενο το παλιό σύστημα όπου είχαμε υποστήριξη της αγοράς και δεν υπήρχε, ε, δεν υπήρχε αστάθεια η διακύμανση των τιμών. Επομένως και ο καταναλωτής είχε μεγαλύτερη σταθερότητα. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα με αυτή την κατάργηση της υποστήριξης των τιμών είναι ότι έχουμε αστάθεια στις τιμές, ε, διακύμανση των τιμών που δεν είναι καλό ούτε για τους καταναλωτές ούτε για τους παραγωγούς. Και αυτό θα μας οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγή σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι καλό για το μέλλον οποιοδήποτε. Και στο τέλος νομίζω ότι θα επανέλθουμε ε, στην αφετηρία, από εκεί που ξεκινήσαμε. Η κυρία τώρα από την Λετωνία έκανε, κάτι πολύ, έκανε κάποιες πολύ καλές παρατηρήσεις για τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και μια μεταβατική περίοδο και πρέπει να, υπάρχει, να λάβουμε υπόψη μας και τις πληρωμές που έγιναν στο παρελθόν διότι δεν μπορείς απλά να κόψεις το σύστημα και να το σταματήσεις χωρίς να αφήσεις μια κάποια λογική μεταβατική περίοδο. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της ΚΟΠΑ. Η κυρία Σαβίνια έχει το λόγο για δύο λεπτά πολύ σύντομα σαν εκπρόσωπο μίας οργανώσεως ε, γεωργών πρέπει να σας πω ότι το πρώτο μέλημα είναι το εισόδημα των γεωργών. Ε, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει εισόδημα γι' αυτό και υπάρχει η δυσαρέσκεια πολλών ε, γεωργών οι οποίοι είναι απογοητευμένοι, έχουν βαρεθεί και περιμένουν να περάσει η μπόρα με φαταλισμό. Ουσιαστικά από τις αρχές του 1990 έχουμε δεχθεί να πληρωνόμαστε σε τιμές που είναι κάτω από το κόστος παραγωγής οπότε χρειάζονται μέτρα ενίσχυσης και οι προτάσεις που διατυπώνουμε αποβλέπουν στην καλύτερη συμβολή στις τιμές αγοράς και γνωρίζουμε ότι ακόμη και από αυτές τις προϋποθέσεις επειδή υπάρχουν διαφορές παραγωγικότητας σε διάφορες περιοχές, ορεινές, πιο δύσκολες θα χρειαστούν υπάρχουν ενισχύσεις και θα παραμείνουν οι ενισχύσεις. Υπάρχει και το θέμα του πλαφών, το οποίο είναι απαραίτητο λόγω της κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν να συσσωρεύονται ε, τόσες ενισχύσεις σε ορισμένους, ενώ άλλοι δεν έχουν τίποτα. Επίσης στη Γεωργία υπάρχει μία αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ γεωργών για αυτό το λόγο. Με, την, ε, ε, με το ανώτατο όριο ορισμένοι αύξησαν τις εκτάσεις τους, κατέστρεψαν τους γείτονές τους και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο και μετά πρέπει να δούμε πώς θα είναι πιο αποδοτικοί οι τρόποι παραγωγής για να ακούμε και τις αγορές και να προωθήσουμε πιο παραγωγικά συστήματα και μια καλύτερη κατανομή σε, σε όλες τις εκτάσεις. Ευχαριστώ. Ο Κοράντο Πίτσο Μπίλο οι περισσότεροι μίλησαν για τις άμεσες πληρωμές, οι οποίες καταρχήν είναι απαραίτητες διότι το 30% είναι ε, από τις άμεσες πληρωμές στο εισόδημά τους και χωρίς αυτές ορισμένοι θα είχαν χρεοκοπήσει. Πολλοί θα είχαν χρεοκοπήσει και δεν θα υπήρχαν τόσα πολλά δημόσια αγωθά, διότι ήδη υπάρχει μία βάση. Χρειαζόμαστε ίσως παραπάνω, αλλά υπάρχει υπάρχει μια βάση. Δεύτερον, όσον αφορά το επίπεδο, πρέπει να μείνει το ίδιο επίπεδο, να αυξηθεί ή να μειωθεί. Πιστεύω ότι πρέπει τουλάχιστον να μείνει στο ίδιο επίπεδο, διότι υπάρχουν νέες αποστολές που έχουν ανατεθεί μέσω της κοινή γεωργικής πολιτικής να αντιμετωπίσουν τις κλιματολογικές αλλαγές, τον ανταγωνισμό στην διατροφική αλυσίδα, τα δημόσια αγαθά και όλα αυτά. Εάν δεν υπάρχει χρηματοδότηση, πώς θα επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι. Και μετά, όσον αφορά τις ε, συνδρομές, την συμβολή. Ε, εμείς διαφωνούμε σε όλα, ε, διαφωνούμε σε όλα τα επίπεδα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Συμβούλιο παντού και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει συμφωνία κατά αυτόν τον τρόπο διότι υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες πάντοτε μπλοκάρουν κάθε απόφαση λέγουν ότι ζημιώνονται πάρα πολύ και κάποιος λέει πρέπει να υπάρχει ένα κατόφλι, ε, κανείς δεν πρέπει να έχει λιγότερο από το 75-80% και αυτό πρέπει να ληφθεί από αυτούς οι οποίοι παίρνουν πολύ περισσότερα στην εθνική βάση και θα δούμε πώς θα τα αναδιοργανώσουμε. Αλλά εγώ δεν βλέπω διαφορετικά πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μην χάνουμε πλέον χρόνο συζητώντας αυτά και ας συζητήσουμε την ουσιαστική μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής πολιτικής που είναι πολύ πιο σημαντική. Σας ευχαριστώ. Ντόουερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νόμιζα ότι είχα δώσει μια σαφή απάντηση σε ένα από τα ερωτήματα και συγκεκριμένα στο πώς μπορούμε να έχουμε ακριβοδίκαιες πληρωμές για τους αγρότες από διαφορετικά κράτη-μέλη. Εγώ είχα πει ότι θα πρέπει αυτό να γίνει σε σχέση με την ε, ε, ισοτιμία αγοραστικής δύναμης σε εθνικό επίπεδο με βάση στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την δυνατότητα, την αγοραστική δύναμη στα κράτη-μέλη είναι ένας δίκαιος τρόπος. Το να περάσουμε σε ισότητα να την Ευρώπη είναι παράλογο όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών στα επίπεδα εισοδήματος αυξάνουν σε μια χώρα τα εισοδήματα, ωφελούνται και οι αγρότες στο πλαίσιο αυτού του 7 ετούς προγράμματος. Τώρα, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές εντός των χωρών. Όχι είναι η απάντησή μου. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα, πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό πάτερν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις άμεσες ε, πληρωμές. Πρώτον, για να περάσουμε, η πρότασή μας ποια είναι για να αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα ε, τις ανισότητες είναι ένα σημαντικό θέμα θα πρέπει να εμείνουμε νομίζω στη χρήση του ε, συνόλου και μετά να δούμε τι θα κάνουμε με τη μετάβαση. Δεν είχα χρόνο να το πω πριν, αλλά αυτό που προτείναμε είναι επιπροσθέτως να υπάρξουν στοχευμένες πληρωμές προς τους αγρότες που προσπαθούν να κάνουν περιβαλλοντικά φιλική γεωργία. Αλλά θα πρέπει να στηριχθούν και να συνεχιστούν να υπάρχουν οι ε, πράσινες ενισχύσεις στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντόουερ. Ο κύριος Σπάν, ο πρόεδρος, έχει Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, όντως η γεωργική πολιτική η κοινή γεωργική πολιτική είναι ένα αποτέλεσμα μιας παράδοσης και αυτό αποτελεί και την αιτιολογία του προτύπου που χρησιμοποιούμε. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν αλλαγές που να συνάδουν με αυτή την ιστορία και όλοι πρέπει να κάνουν περαιτέρω ε, προτάσεις για να προχωρήσουμε. Αλλάζει η γεωργία, αλλάζει η κοινωνία και ως εκ τούτου και η αιτιολογία και η χρήση αυτών των μέσων πρέπει να ξανααιτιολογηθεί και γι' αυτό είναι σωστές οι προτάσεις του Επιτρόπου ε, και γι' αυτό τη στηρίζουμε. Σήμερα υπάρχει μια κατάσταση όπου πλέον το πρόβλημα δεν είναι ε, αν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την προμήθεια τροφίμων στην Ευρώπη αλλά να υπάρξουν και νέες μέθοδοι και γι' αυτό ζητούμε το θέμα της απασχόλησης να αποτελέσει ένα στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να αντικατοπτρίζεται στην κοινή γεωργική πολιτική. Αυτό πρέπει να συζητηθεί το 2001 όχι με περιορισμούς αλλά με ανοιχτές πόρτες και κατανόηση. Πρέπει να υπάρχει και δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν πρέπει όλοι να έχουν τα ίδια διότι αυτό το πρότυπο έχει αποτύχει αλλά ο καθένας θα πρέπει να βρίσκει τη θέση του σε αυτό το ευρωπαϊκό κοινό οικοδόμημα και είναι πολύ βασικό να συζητήσουμε ποιες παραμέτρους θα χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιήσουμε εάν θα πάρουμε το μέσο όρο του εθνικού εισοδήματος, του κοινοτικού εισοδήματος θα πρέπει να καθίσουμε και να συνεννοηθούμε, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και ε, ίσως ε, να θεωρήσουμε ότι οποιοδήποτε ανώτατο επίπεδο κάτω από τα 3.000 ευρώ θα χρεοκοπούσε ε, τα νοικοκυριά των γεωργών και πρέπει να υπάρχει μια βιώσιμη ανάπτυξη και όχι καταστροφή για τους γεωργιούς. Ευχαριστώ. Η τελευταία ομιλήτρια η κυρία Μέλλον είναι δύσκολο να απαντήσω σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σε όλες τι ερωτήσεις. Να θίξω κάποια με σημαντικά θέματα όμως. Το τελευταίο σχόλιο που έγινε για την ε, ΚΑΠΑ που δεν είναι μια ε, κοινωνική υπερβολοντική πολιτική αλλά είναι μια γεωργική πολιτική. Εμείς πιστεύουμε ε, ότι δεν θα πρέπει να χωρίζουμε την πολιτική αυτή σε ε, διάφορους τομείς. Ε, αυτό που μετράει είναι να έχουμε μια συνεκτική πολιτική. Δεν μπορεί να κρατήσει η πολιτική αυτή και να σταθεί εάν απευθύνεται μόνο σε ένα κομμάτι του, πάνελ, του πάζλ. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε στα διατροφική αλυσίδα είναι να είναι μια συνεκτική ε, αντιμετώπιση. Υπάρχουν πολλές πολιτικές προφανώς και όταν είσαι στη μέση και προσπαθείς ε, να τις εφαρμόσεις όλους και να σεβαστείς όλους τους κανόνες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως, ναι, λέμε ότι όντως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον, ε, και τον ε, κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό πυλώνα της βιωσιμότητας. Τώρα, επανεθνικοποίηση όχι, δεν θέλουμε. Δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θέλουμε μια προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης για την ερώτησή σας κύριε Μποβέ αναφερθήκατε στις πληρωμές που θα στηρίζονται στην παραγωγή. Ε, που συνδέονται με το κόστος παραγωγής. Ε, το συζητήσαμε με, και πρέπει να το συζητήσουμε και με τους ε, υπεύθυνους του λιανεμπορίου. πρέπει να δούμε όλη την αλυσίδα δηλαδή. Αυτό είναι ένα από τα καθήκοντα του φόρουμ υψηλού επίπεδου. Θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα και ίσως θα μπορούσαμε στο φόρουμ ανταγωνιστικότητας της διατροφικής αλυσίδας να το συζητήσουμε. Ε, αν θέλετε μετά την συνεδρίαση αυτή μπορούμε να σας, δώσουμε, να σας ενημερώσουμε για τις ιδέες που έχουμε εμείς σαν κλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε πολύ προσεκτικοί και με το χρόνο. Μας περνάμε στη δεύτερη συνεδρία που αφορά τα μέτρα της αγοράς. Θα διαβάσω τον κατάλογο των τριών ερωτήσεων και θα ζητήσω από το πάνελ να απαντήσει χωρίς να ξεπεράσουμε τα τρία λεπτά. Αυτή τη φορά το... δεν έχουμε τον ε, πρόεδρο της ΚΟΠΑ, έχουμε τον πρόεδρο της ΚΟΖΕΚΑ, τον κύριο Μπρούνι. Λοιπόν, η ερωτήση είναι η ποιες σχέσεις υπάρχουν ανάμεσα στην, ε, στα μέτρα της αγοράς και της, ε, πολιτι... της ε, πολιτικές για το διεθνές εμπόριο δεύτερη ερώτηση, είναι εφικτό να αντικαταστήσουμε τη, τα υπάρχοντα δίκτυα ασφάλειας ε, της αγοράς ε, με το προτινόμενο, εργαλείο, με την προτινόμενη εργαλειοθήκη, αν θέλετε, για διαχείριση των κινδύνων και ποια μέτρα είναι απαραίτητα ε, για να μπορέσουν οι παραγωγοί να εξασφαλίσουν ένα δίκαιο εισόδημα. Πρώτη ομιλήτρια το να δημιουργηθούν αυτά τα εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ε, αντιμετωπίσουμε τη διακύμανση των διαφόρων ε, στοιχείων ε, από τις οποίες εξαρτάται η παραγωγή και η παραγωγή και με όμικρον και με γιώτα, δηλαδή ας πούμε διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών κτλ. Θα πρέπει να μπορέσουμε να επίσης ε, να έχουμε στη διάθεσή μας κάποια εργαλεία τα οποία θα ε, αντισταθμίσουν κάπως την διακύμαση της αγοράς τονίζουμε την ανάγκη να υπάρχει παραλληλισμός με την ε, κατάργηση των ε, ε, ενισχύσεων για τις εξαγωγές ούτως ή άλλως σύμφωνα με τον ΠΟΕ για την κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων θα πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα και κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζουν παράλληλα τα κράτη-μέλη. Εμείς θεωρούμε ότι πάρα πολλά εργαλεία ε, μας επιτρέπουν να αποφύγουμε τις κρίσεις. Δεν συμφωνούμε με όλο τον κατάλογο, αλλά να σας δώσω κάποια παραδείγματα ε, για την τα εργαλεία για την διαχείριση των κινδύνων. Τα συζητήσαμε Μπορούν να βοηθήσουμε τους παραγωγούς για να αντιμετωπίσουν κάποιους κινδύνους που οδηγούν στην βιωσιμότητα της γεωργικής κοινότητας. Σαν κομμάτι του δεύτερου πυλώνα πρέπει να είναι συμβατά με τον ΠΟΕ. Εξετάσαμε και τις μελλοντικές αγορές που θα βοηθήσουν ε, ε, τους ε, παραγωγούς να περιορίσουν την διακύμανση των τιμών και να προστατευτούν από αυτή τη διακύμανση. Η Κομισιόν θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη χρήση τους, ενημερώνοντας καλύτερα τους ενδιαφερομένους. <laughs> Αν νόμιζα ότι μου γνέφατε και νόμιζα ότι πέρασα τον χρόνο μου. Τώρα για το τελευταίο ερώτημα. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα κάποια εργαλεία που αφορούν την αγορά, κάποια δίκτυα ασφαλείας, ή ε, ε, αγορές ε, για τα παράγωγα προϊόντα. Επίσης υπάρχουν και εργαλεία που ανήκουν στο δεύτερο πυλώνα που μπορούν να βελτιώσουν την αγωνιστικότητα του κλάδου, επενδύσεις, ενισχύσεις για επενδύσεις και για καινοτομία, βελτίωση της γνώσης, βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού. Ε, ποιοτικά μέτρα και βοήθεια για την απόκτηση προσόντων, περισσότερων προσόντων. Τέλος πάντων, υπάρχουν μια, υπάρχει μια σειρά μέτρων και εργαλείων που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ο πρόεδρος Μπρούνι της Κοζέκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Στην προηγούμενη συνεδρία παρενέβη ο πρόεδρος της ΚΟΠΑ. Εγώ είμαι πρόεδρος της ΚΟΖΕΚΑ. 38.000 ε, συνεταιρισμοί στην Ευρώπη. Ε, έχουμε με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε δισεκατομμύρια. Θα ήθελα να επαντήσω στις ερωτήσεις σας ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και για την δυνατότητα που μας δίνεται να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πρώτη ερώτηση που αφορά τις, τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να το εξετάσουμε, να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τις διεθνείς πολιτικές. Κάθε παραχώρηση ε, που γίνεται σημαίνει μεγαλύτερα προβλήματα για τους παραγωγούς. Δείτε τι έγινε στην, με τη Μερκοσούρ και το Μαρόκο. Οι συμφωνίες αυτές ε, ε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ευρωπαίους παραγωγούς. Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν όλοι οι κανόνες για τα ποιοτικά πρότυπα, τα οποία δεν είναι ίδια με αυτά τα οποία ε, επιβάλλονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ε, υπάρχει και πρέπει να τονίσουμε μια μεγάλη πρωτοβουλία που ξεκίνησε το Κοινοβούλιο πέρσι τον Ιούλιο και αφορά την ε, επισήμανση για την προέλευση και εδώ όμως έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες από πλευράς του Συμβουλίου των Υπουργών Υγείας είχαμε μια υπαναχώρηση γι' αυτό ακριβώς θέλουμε το Κοινοβούλιο να ξεκινήσει ξανά το θέμα της ε, σήμανσης προέλευσης το, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να α, ε, διαφυλάξουμε τη γεωργία στην Ευρώπη σημαίνει ε, να διαφυλάξουμε και την απασχόληση. Έχουμε 7 εκατομμύρια ακούστηκε γεωργούς, όμως ε, αυτή εγώ πιστεύω ότι ένα στου έξι εργαζόμενους στην, στην Ευρώπη εξαρτάται από τον γεωργικό τομέα. Επομένως, είναι ζωτική σημασία να διαφυλάξουμε την γεωργία. Ε, δεύτερη ερώτηση που αφορά την αντικατάσταση των δικτύων δικτύων ασφάλεια, ε, με κάποια άλλα εργαλεία. Θυμηθείτε τι έγινε πέρυσι με τα δημητριακά, με το γάλα κτλ. Δι, δι, βλέπετε ε, ποιοι είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η γεωργία, κίνδυνους που προέρχονται από την αγορά. Τώρα, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πιο δίκαιο εισόδημα. Εδώ θα πρέπει να ε, ε, επανασορροπήσουμε τη διατροφική αλυσίδα, διότι όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν στη διατροφική αλυσίδα δεν συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο, δεν έχουν τις ίδιες ε, υποχρεώσεις. Η παραγωγή είναι, αν θέλετε, προωθούν την, ε, και μεταφέρουν την εκμετάλλευση, την, ε, την πρόσβαση της εκμετάλλευση στην αγορά. αυτή, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Ιουμπρούνη. Η κυρία Σαβίνια έχει το λόγο. Σαβινή, πάμε. Το θέμα των εργαλείων της αγοράς, των ε, μέτρων της αγοράς, νομίζουμε ότι είναι το επίκεντρο αυτής της τέταρτης επιλογής που προτείνουμε εμείς. Είναι σημαντικό, ακόμη κι αν είναι πολύ κεφαλαίο σημασία βέβαια οι ενισχύσει, ότι ο, ο των εκμεταλλεύσεων κατά 50, 60, 80 ή 100% ε, σε κάποιες παραγωγές και σε κάποιες χώρες εξαρτάται από την πώληση προϊόντων. Άρα το θέμα της τιμής είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξασφάλιση του εισοδήματος και πρέπει να το έχουμε συνέχεια υπόψη μας. Η Κομισιόν συχνά μιλά για δίκτυα ασφαλείας. Εμείς νομίζουμε ότι είναι σημαντικότερο να μιλάμε για μια εργαλειοθήκη που ως το δυνατόν περισσότερα εργαλεία θα έχει για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα όσα συμβαίνουν σήμερα και δι' αυτές τις ε, διακυμάνσεις που δημιουργούν τόσα προβλήματα. Μεταξύ αυτών των εργαλείων νομίζουμε ότι τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων που προτείνει η Κομισιόν δεν είναι καλά εργαλεία είναι σαν να βάζει σε σελοτέιπ ε, σε, μια, ε, σε κάτι που έχει σπάσει. Δεν ε, αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, ε, τα θέματα, τα προβλήματα που τίθενται. Εξού λοιπόν και όταν τελικά οι αγορές κατακλειστούν από κερδοσκόπους παράγοντες δεν μπορούν να φέρουν τη σταθερότητα που είναι ευκταία. Το ίδιο ισχύει και για τις ασφάλειες σε σχέση με τα, με τα υγειονομικά προβλήματα ή το κλίμα. Εκεί μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, αλλά όταν μιλάμε για το εισόδημα που σχετίζεται και με άλλα θέματα, φυσικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα διακυβεύματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν καλά εργαλεία στην εργαλειοθήκη, που κάποια από αυτά είναι παλιά, αλλά πρέπει να τα συντηρήσουμε ώστε αν χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε. Και βέβαια θα υπάρχει έτσι και ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες. Μεταξύ των εργαλείων αυτών νομίζω ότι μπορούμε να επιμείνουμε σε κάποια που μας φαίνονται σημαντικά. Έλεγχος παραγωγών. Παραγωγών ή υποπαραγωγών στο θηλυκό μυλό. Σε ό,τι αφορά και την εξαγωγική ικανότητα για να μην υπάρχει ανάγκη επιδοτήσεων. Γαλακτοκομικές ποσοστώσεις που φέρανε μεγάλη σταθερότητα στην αγορά του γάλακτος για πολλά χρόνια. Αποθέματα επίσης, στρατηγικά αποθέματα για, τα δημητριακά, για τις παραγωγές δημητριακών μπορούν να φέρουν σταθερότητα και επιστηστική ασφάλεια. Και νομίζω ότι σήμερα είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας όταν η διεθνής αστάθεια δημιουργεί σοβαρές κρίσεις μεταξύ αυτών και Σοβαρέ πολιτικές κρίσεις. Ως Ευρωπαίοι πολίτε, νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη. Εργαλεία που έχουν αποδείξει την αξία τους δεν πρέπει να τα πετάξουμε, αλλά να τα αξιοποιήσουμε στους επόμενους μήνες. Ο κύριος... Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάννα για τρία λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η διεθνής ε, εμπορική πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί και στην ε, Ευρώπη αλλά θα πρέπει να ισχύσει στην Ευρώπη και η διεθνής νομοθεσία για την ε, διατροφική ασφάλεια και θα πρέπει καταρχήν να μπορούμε να τροφοδοτούμε τον πληθυσμό της Ευρώπης και μετά να εξάγουμε αλλά αυτό χρειάζεται μια μεγάλη συζήτηση διότι θα χρειαστούν και εξαγωγικές ενισχύσεις και ε, για να ε, μπορέσουμε να αντιταχθούμε σε άλλα γεωργικά κράτη. Βλέπουμε ε, ότι ορισμένες βιομηχανίες συγκρίνουν ε, με τη βιομηχανία που μπορεί να μετατοπίσει μία παραγωγή για το επόμενο έτος ενώ πρέπει να φάμε κάθε μέρα. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να υπάρχει ήδη αντιμετώπιση διότι πιστεύω ότι αυτό είναι τα μία ε, αντιμετώπιση ιδεολογική και στο μέλλον πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν πολυμερείς λύσεις οι οποίες δεν πρέπει όμως να είναι καταστροφικές. Αυτοί οι οποίοι μας δίνουν αυτά τα νέα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο είναι αυτοί οι οποίοι συμβάλλουν στην καταστροφή μας. Εμείς δεν, δεν είμαστε ενάντια στην ύπαρξη νέων μέσων αλλά πρέπει να έχουν αξιολογηθεί πράγμα που δεν έχει γίνει στο παρελθόν και ελπίζουμε ότι αυτή η Επιτροπή θα διατηρήσει τα ισχύοντα μέτρα μέχρι ότου υπάρξουν οι αποδείσεις για τα νέα μέτρα όπως άλλωστε είπε και ο κύριος Γουόλς από την, ε, ε, Κόπα. Ε, τώρα, τι μπορούμε εμείς να ζητήσουμε. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των τιμών της διατροφικής αλωσίδας που ξεκίνησε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση των τιμών στην Ευρώπη και ε, παρόλα αυτά ε, έχουμε μετατοπίσει την, ε, τις παροχές υπηρεσιών που χρειάζεται η γεωργία για να παράγει και αυτό είχε δραματικές επιπτώσεις διότι δεν έχει ενισχύσει τους ε, ε, τους γεωργούς μας και δεν μπορεί να συμβάλλει σε μία λογική διαμόρφωση τιμών. Βλέπουμε ότι αν συγκρίνουμε τους μισθούς με τις άλλες βιομηχανίες υστερούμε και γι' αυτό δεν έχουμε ειδικευμένο εργατικό προσωπικό. Χρειαζόμαστε νέες δυνατότητες. Δεν είναι δυνατόν τώρα να λύσουμε το θέμα αυτό στα πλαίσια της γεωργικής πολιτικής αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστεί επίσης να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Πίτσο Βίλιο. σχετικά με το πρώτο θέμα ε, όσον αφορά ε, τις ε, εμπορικές σχέσεις. Πιστεύουμε ότι πρέπει να μπορέσουμε καταρχήν να σεβαστούμε τις αρχές του ΠΟΕ αλλά συγχρόνως να προστατεύσουμε την παραγωγή μας. Άρα το ερώτημά μας δεν είναι αν συνάδει η κοινή γεωργική πολιτική με το διεθνές εμπόριο αλλά αν το διεθνές διεθνές εμπόριο συνάδει με την πολιτική μας και όπως είπαν ήδη ορισμένοι θα πρέπει να υπάρξουν νέες ε, ε, ε, θα πρέπει να, δεν θα πρέπει να υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις με τις χώρες του Μερκοσούρ διότι η κίνηση αυτή είναι ανεύθυνη. Όσον αφορά τα μέσα τα οποία πρέπει να διατεθούν όπως είπαμε Υπάρχουν νέες δυνατότητες μέσω των νέων μέτρων αλλά και μεγαλύτερη ε, αστάθεια και το βασικό θέμα είναι εάν μπορούμε να επέμβουμε για ορισμένες πρώτες ύλες. Ε, το πρόβλημα όμως παραμένει όσο διατηρούνται υψηλές τιμές και ε, η επέμβαση για το γάλα ίσως αποδίδει αλλά σε άλλους τομείς δεν έχουμε αποτελέσματα όταν υπάρχουν μέσα σταθεροποίησης τιμών και αλλού ή όταν δεν υπάρχουν. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι οι άμεσες πληρωμές είναι ο καλύτερος τρόπος για να σταθεροποιήσουμε το γεωργικό εισόδημα στην Ευρώπη και ε, θα απαντούσα όσον αφορά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, μία σωστή ανταμοιβή για την παραγωγή ότι θα χρειαστεί συνεργασία των γεωργών και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχουμε ένα χρηματιστήριο των ε, πρώτων υλών για μελλοντικές αγορές όπως το Σικάγο και στην Ευρώπη. Αναφέρω αναφέρομαι και στην ε, έκθεση Μποβέ, η οποία είναι ουσιαστική και με οδηγεί στο τελευταίο θέμα. Εάν ανταμείβουμε δηλαδή σωστά τους ε, γεωργούς οι οποίοι έχουν ε, ελάχιστο ποσοστό ε, του συνολικού κόστους που καταβάλει ο καταναλωτής από 50% βρισκόμαστε στο 10-15% και θεωρώ ότι η έκθεση Μποβέ είτε είναι η πιο ουσιαστική εισήγηση η οποία καταρτίστηκε τον τελευταίο καιρό. Ευχαριστώ και τώρα ο τελευταίος είναι ο κύριος Ντόουερ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τη Βία Καμπεσίνα. Πρέπει οι αγρότες να έχουν δίκαια καλή απόδοση. Γιατί αν δεν το καταφέρουμε αυτό θα δαπανούμε όλους τους πόρους των φορολογουμένων για αύξηση του εισοδήματο των αγροτών. Άρα πρέπει να γίνουν προσπάθειες και δικαιολογούνται κάποιες δαπάνες για να υπάρχουν αυτά τα αυτή η δίκαιη απόδοση. Δύο μέτρα θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν. Πρώτον, στήριξη και ίσως και αλλαγή του ε, νόμου περιεταγωνισμού ώστε να μπορούν να δημιουργούν οι αγρότες κάποιες ομάδες εμπορίας για να αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη και να μπορούν να διχειριστούν την ε, προσφορά και να προσθέσουν αξία ή δυνατόν στα προϊόντα τους. Τονίζω ότι μιλάμε για ομίλους που ελέγχονται από τους αγρότες, όχι από αγρότες και άλλους στο πλαίσιο της διατροφικής αλυσίδας όπως συμβαίνει με κάποιους συνεταιρισμούς. Δεύτερον, δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Παρακολούθησης των Αγορών που θα έχει τα εξή καθήκοντα. Συνεχή παρακολούθηση της κίνησης τιμών, κόστος παραγωγής, προσφορά ζήτησης. Βάση του κόστος παραγωγής, καθορισμός ενός διαδρόμου τιμών για κάποια προϊόντα, μιας περιοχής τιμών. Και όταν οι τιμές υπερβαίνουν ή είναι πολύ χαμηλότερες αυτού της περιοχής τιμών, αύξηση ή μείωση παραγωγής. Και όταν υπάρχει σημαντική υπερπαραγωγή, άρα μειώνονται σημαντικά οι περιοχές, οι τιμές, αγορά περιορισμένων μετοχών ή αποθεμάτων με τη χρήση πόρων που εισπράττονται από όλου του σχετικού παραγωγού. Για τα άλλα θέματα, κατά την άποψή μας, τα εφισταμένα δίχτυα ασφάλειας δεν θα πετύχουν τους στόχους αυτούς, γιατί είναι πολύ χαμηλές τιμέ παρέμβασης. Η ασφάλεια δεν είναι λογική λύση και ούτε σταθεροποιούνται οι τιμέ μέσω των αγορών παραγόγων. Και σε ό,τι αφορά το εμπόριο, οι κακέ εμπορικέ πολιτικέ μπορούν να να καταστρέψουν αυτά τα οποία μπορούν να φτιάξουν οι καλοί κανονισμοί για το εμπόριο. Άρα δεν πρέπει να επιδοτούμε τις εξαγωγές τροφίμων. Πρέπει να διαχωρίσουμε τη Γεωργία από άλλους κλάδους ε, στις παγκόσμιες εμπορικές ε, συζητήσεις όπως Μερκοσούρ για παράδειγμα και να επιμείνουμε ότι πρέπει να υπάρχουν ε, τα ίδια πρότυπα για τις εξαγωγές τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά που ισχύουν για το εντός της Ένωσης τρόφιμων. Ευχαριστώ όλους. Περνάμε τώρα στο, στη στο δεύτερο κομμάτι της ε, συνεδρίας, αν θέλετε, όπου έχουμε εννέα ομιλητές από, την, ε, από, τα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να ε, ε, πείτε σε ποιον απευθύνεται την ερώτηση. Η πρώτη Ομιλήτρια είναι η Μέριντ Μαγκίνες. Ευχαριστώ τον, ε, το πάνελ. Απαντήσανε πάρα πολύ καλά. Πρώτη ερώτηση στον πρόεδρο της ΕΛΟ. Εάν ε, είναι η στάση της Κομισιόν απαράδεκτη ε, όσον αφορά τις συμφωνίες με, το, με τη Μερκοσούρ και το Μαρόκο, γιατί γίνεται αυτό. Επίσης έχουμε την παραδοσιακή παρα, παρέμβαση και την ε, αποθεμα, αποθεματοποίηση που είχαμε τότε. Εάν έπρεπε να επιλέξουμε τα παλιά εργαλεία που είχαμε και τα καινούργια ε, εργαλεία τα οποία τώρα προτείνονται, εσείς με ποια θα αισθανόσαστε πιο άνετα. Τώρα όσον αφορά την αλυσίδα προμήθειας, η πρώτη παρέμβαση αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, η κυρία Φρούεν. Όμως θα ήθελα να ακούσω λίγο παραπάνω για την λύση. Γιατί πιστεύουμε ότι αν δώσουμε μεγαλύτερη δύναμη στους παραγωγούς μέσα στα πλαίσια των ομάδων παραγωγών, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Επίσης, θα ήθελα να σας ζητήσω να σχολιάσετε τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία και πώς ε, η υποστήριξη της αγοράς απαιτείται για να γίνει αυτό με βάση τις απαιτήσει μας για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ε, ερωτήματα. Επίσης, η ερώτησή μου αφορά το παρελθόν τώρα η τελευταία η Κομισιόν ήθελε να, να εξαφανίσει τα μέτρα που υποστήριζαν την αγορά, διότι θεωρούσαμε ότι η αγορά ήταν... πήγαινε καλά. Πιστεύετε ότι ίσως προχωρήσαμε πάρα πολύ όσον αφορά το δίκτυο ασφαλείας και θα έπρεπε να έχουμε κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ την Μάια. Κασία Περές. Ευχαριστώ πολύ. Αν στην πρώτη συζήτηση, στην προηγούμενη συνεδρία, συμφωνήσαμε ότι είναι σημαντικές οι άμεσες πληρωμές, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και εδώ ότι παρά τα αυτά δεν μπορούμε χωρίς άμεσες πληρωμές να εγγυηθούμε τη βιωσιμότητα του τομέα. Αν δεν μπορέσουμε να ενσωματώσουμε εργαλεία διαχείρισης των αγορών, που όπως άκουσα και από μία άλλη ε, προλαλήσασα, τα ε, ξεφορτωθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και τώρα βλέπουμε ότι πρέπει να ενσωματώσουμε κάποια από αυτά τα εργαλεία και πάλι για να αγγιθούμε δίκαιες τιμές αλλά να αγγιθούμε και το εισόδημα των αγροτών. Το θέμα των ταμείων, ε, το θέμα της διακύμασης των τιμών των πρώτων υλών το βλέπουμε σε τομείς όπως αυτός της κτηνοτροφίας σήμερα. Πολλές φορές επίσης βλέπουμε ότι καθυστερεί και λήψη αποφάσεων θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε σε αυτή τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής να ενσωματωθούν και κάποιοι μηχανισμοί έγκαιρης αντίδρασης των ευρωπαϊκών αρχών σε συγκεκριμένα προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζει σήμερα η κτηνοτροφία. Κατά το παρελθόν ε, ο γαλακτοκομικός τομέας είναι σημαντικό να δίνεται μια ταχύα απάντηση από τις κοινοτικέ αρχές. Και τέλος, ε, φαντάζομαι θα συμφωνήσουν μαζί μου και οι συγκητές, ένα θεμελιώδες ζήτημα είναι η αμοιβαιότητα. Έγινε μνήμα σε αυτήν και θα πρέπει να είμαστε σε θέση σε αυτή τη μεταρρύθμιση να συμπεριλάβουμε και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αμοιβαιότητα. Γιατί καλό είναι να αυξήσουμε τα ποιοτικά πρότυπα των προϊόντων μας και τις καλή μεταχείρισεις των ζώων, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να μπορούμε να απαιτούμε τις απαιτήσει αυτές, να τις πληρούν και τρίτα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. James Nicholson έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ το πάνελ. Είναι πολύ δύσκολος ο τομέας. Υπάρχουν πολλές ιδέες. Το πρόβλημα με τις ιδέες είναι, όταν υπάρχουν πολλές ιδέες, είναι ποιες είναι από αυτές που θα είναι αποτελεσματικές. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Μιλήσαμε για διακύμανση των τιμών. Ε, τι στα σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι, ε, και βλέπουμε ε, τα σούπερ μάρκετ δεν βγάζουν λεφτά, οι ενδιάμεσοι δεν βγάζουν λεφτά, οι παραγωγοί δεν βγάζουν λεφτά. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς στην Ευρώπη λέμε ότι έχουμε τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής, ε, φροντίζουμε για τα ζώα κτλ. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται με τα τρόφιμα τα οποία εισάγονται στην Ευρώπη, που δεν πληρούν ε, τα στάνταρ τα οποία είναι υποχρεωμένοι οι παραγωγοί μας να σεβαστούν. Πιστεύουμε ότι πρέπει να, ότι πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας. Δίδατε και στην προηγούμενη κρίση τι έγινε. Μονάχα όταν εισάγαμε αυτό το δίκτυο ασφαλείας ε, διορθώθηκε η κατάσταση. Εύκολα πηγαίνανε τα, τα τρόφιμα στην παρέμβαση και μετά, στην αποθεματοποίηση συγγνώμη, και μετά α, πάρα πολύ εύκολα και με καλό κέρδος πουλήθηκαν τα προϊόντα που ήταν στην αποθεματοποίηση. Δεν ξέρω, μήπως θα μπορούσαμε να, τα, να το δούμε αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά. Είδαμε τον, τι γίνεται και στον, και στον ΠΟΕ. Είδαμε επίση τι γίνεται και με τι διμερεί συμφωνίε όπω με την Μερκοσούρ. Όλοι μα λένε ότι πρέπει να παράγουμε περισσότερο φαγητό, περισσότερο τρόφιμα. Αλλά πώ όμω μπορούμε να ζητήσουμε από του παραγωγού μα να παράγουν περισσότερα τρόφιμα με λιγότερε και λιγότερες, λιγότερα έσοδα. Κύριος Φοντάνα, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν εδώ σήμερα και, για να μας απαντήσουν. Ε, ε, οφείλω να ομολογήσω ότι έχω πάρα πολλά κοινά με τον προλαλήσοντα, τον κύριο Νίκολσον, γιατί οι ερωτήσεις είναι ίδιες. Όντως υπάρχει αυτή η διακύμανση των τιμών που οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλά τρόφιμα τα οποία προέρχονται, εισάγονται στην κοινότητα ε, με χαμηλό κόστος, δεν έχουν την ίδια ποιότητα με τα δικά μας και δεν έχουν παραχθεί σεβόμενοι τις περιβαλλοντικές ε, επιταγές. Και θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω τι πιστεύετε για αυτό το θέμα. Γιατί τα, μήπως έπρεπε τα προϊόντα τα οποία εισάγονται στην ε, κοινότητα να σέβονται τα ποιοτικά κριτήρια και τα παραβολητικά κριτήρια τα οποία ε, επιβάλλουμε στην εγχώρια παραγωγή. Μάλλον θα συμφωνείτε βέβαια. Μια άλλη ερώτηση. Ένα τμήμα της Επιτροπής διστάζει η Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάω, για τη στάση να αντιμετωπίσει το θέμα των εμπορικών συναλλαγών, των διεθνών συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια της ΚΑΠ. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς το βλέπετε εσείς αυτό, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα για να μπορούν οι παραγωγοί μας να παράγουν ανταγωνιστικά μέσα σε ένα περιβάλλον αθέμη του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ Λορέντσο, η Ελίζα Πεθιέγγελη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ ε, θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους εισηγητές και χαίρομαι ότι συμφωνήσαμε στον πρώτο γύρο ότι πρέπει να χρειαστεί ένας ισχυρός πρώτος πυλώνας. Αυτό που δεν άκουσα στον πρώτο γύρο ήταν ε, ο έλεγχος ε, για το, εντός του πρώτου πυλώνα, το screening, ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Όσον αφορά τα μέτρα της αγοράς, πρέπει να σας πω ότι συμφώνησα με αυτά που είπε στην αρχή η Κοπάκο Ζεκά. Θα ήθελα όμως να τους ρωτήσω μήπως ε, κάναμε υπερβολική απελευθέρωση ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως ε, προχώρησε υπερβολικά και τι θα έπρεπε να συνεχίσουν να υπάρξουν σαν μέτρα στην αγορά, προστασίας αγοράς σαν δίχτυ ασφαλείας διότι θεωρώ ότι ε, ε, ε, υπάρχει ένα θέμα για την επιβίωση. Εσείς γιατί απορρίπτετε την αναπτυξιακή βοήθεια διότι για να επιβιώσουμε πιστεύω ότι τη χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη αλλά θα ήθελα να το σχολιάσουν και οι άλλοι συγγητές. Όσον αφορά την ε, ε, εμπορική πολιτική και εγώ συμφωνώ ότι κάθε παραχώρηση μας δημιουργεί προβλήματα. Τι λοιπόν θα είναι η δικιά σας θέση ε, για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό μέσα μέτρα στην αγορά διότι στην Ευρώπη έχουμε τις ύψιστες προδιαγραφές για την υγιεινή των τροφίμων και ούτω καθεξής. Άρα και εκεί πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε διότι μας λέτε ότι έχουμε εξασφαλίσει την ελάχιστη τροφοδότησή μας αλλά βλέπετε πόσο γρήγορα μπορεί να υπάρξει πρόβλημα εάν κάτι προκύψει και πόσο σημαντική και εξασφαλισμένη είναι η κυριαρχία μας γιατί είπατε ότι όταν τα τρόφιμα ε, γίνονται πάρα πολύ ακριβά υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ε, ε, διεκόπησε την ομιλήτρια. Ο κύριος Παύλο Χάλτες για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Κάθε προϊόν της αγοράς έχει τα ίδια χαρακτηριστικά του, έχει ρυθμιστικούς μηχανισμούς για να μην έχουμε ε, απότομες αυξομοιώσεις στην αγορά, ε, στις τιμές και στην αγορά ε, και το θέμα της διαμορφώσεως των τιμών υπερβαίνει το τομέα της γεωργίας αναφέρεται και στον ανταγωνισμό και τα δημοσιονομικά μέτρα και εξαρτάται και από άλλους οργανισμούς όπως είναι το G20. Επηρεάζονται όμως οι γεωργοί οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίσουν επαρκή παραγωγή τροφίμων για την Ευρώπη αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις διαστάσεις της γεωργίας. Όσον αφορά την μεταρρύθμιση της ε, ε, γεωργικής πολιτικής και την επίτευξη των στόχων της μπορεί αυτό να γίνει μόνο ε, εάν μπορέσουμε να εμπλέξουμε και τις άλλες πολιτικές διότι όταν μιλάμε για τα εισοδήματα, πρέπει ε, να σκεφτούμε τις, ε, ε, τις δημοσιονομικές κρίσεις και δεν πρέπει να διαταράσουμε την διατροφική αλυσίδα. Έχουμε όμως προβλήματα με τους διανομής και αν όταν εξετάζετε τις αυξήσεις των τιμών βλέπετε ότι μπορεί μεταξύ της παραγωγής και της διάθεσης υπάρχει μία αύξηση κατά 50% για την οποία ευθύνονται κατά πολύ διανομής. Μήπως λοιπόν πρέπει να γίνει μία ανακατάταξη διότι τελικά δεν έχουμε να προσφέρουμε σωστές λύσεις. Η... Ε, διεκόπη ο μιλητής. Μισελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους, ε, τα μέλη του πάνελ. Όταν μιλάμε για κοινή γεωργική πολιτική, μιλάμε για διατροφικούς πόρους. Όταν μιλάμε για κάπα, μιλάμε για προϊόντα κατανάλωσης. Ε, είμαστε εδώ στον πυρήνα της κοινή γεωργικής πολιτικής και αυτό διότι θέλουμε να διαχειριστούμε τους διατροφικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ούτως ή άλλως τα αιτήματα για τρόφιμα αυξάνουν κατά 3% κάθε χρόνο. Ενώ η αγορά αυτή, ο κλάδος αυτός συρρυκνώνεται συνέχεια. Τα, ένα μεγάλο, μεγάλο μέρος των γεωργικών προϊόντων ε, τίθεται σε εμπορία στην ε, περιοχή όπου παρήχθησε. Και ρωτώ, θα έπρεπε όπως ε, προβλέπουν ή ζητάνε κάποιοι να εφαρμόσουμε μια διπλή πολιτική που κάνει διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτά τα οποία παράγονται και κυκλοφορούν στην περιοχή που παρήχθησαν και σε σχέση με τα υπόλοιπα τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο εκτός της περιοχής παραγωγής. Δεύτερον, πώς μπορούμε να θέσουμε σε εμπορία τα αποθέματα και πώς μπορούμε να τα πληρώσουμε. Και τρίτο ερώτημα που απευθύνεται στον εκπρόσωπο του Άρκο 2020. Είπατε ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση όταν αυξάνονται οι τιμές να αυξάνουμε την παραγωγή και όταν μειώνονται οι τιμές να μειώνουμε την παραγωγή. Γεωργία χρειάζονται εννέα μήνες, ένα χρόνο ή ίσως και τρία χρόνια για να δημιουργηθεί ένα εργαλείο παραγωγής. Επομένως εσείς πώς βλέπετε να ισχύουν όλα αυτά τα οποία είπατε. John Stuart Agnew, δύο λεπτά. Συμφωνεί το πάνελ ότι σε ένα χρόνο εάν δεν έχουμε μία μια σωστή μεταρρύθμιση ο παραγωγός αυγών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα μπορεί να ανταγωνιστεί σωστά τους υπόλοιπους παραγωγούς. Οι χώρες που δεν συμμορφώνουν, δεν, που δεν έχουν συμμορφωθεί δεν μπορούν να... δεν θα μπορέσουν δεν θα, δεν θα, πρέπει, να, δεν θα πρέπει να υποφεληθούν από τα πλεονεκτήματα και αυτά τα κράτη ε, ε, που, που επιτρέπουν την παραγωγή αυτών των αυγών θα πρέπει να τα σημαδέψουν αυτά τα αυγά και θα πρέπει να, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Τέλος πάντων, ήθελα να πω επίσης ε, για την Gyrotech που είναι μια ε, ουγγρική εταιρεία ε, η οποία έχει σαν στόχο να βελτιώσει την ευζοία των σκύλων. Δόθηκαν χρήματα σε αυτή την εταιρεία και ε, τελικά δεν, έγιναν, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Απλώ αγοράστηκαν γραφεία, προσελήθη προσωπικό και, και οι επενδυτέ ανησυχούν και τα ουγγρικά σκυλιά επίση. Ο κύριος Γκουτιέρες. Ευχαριστώ Πάολο, συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπες. Η τάση η οποία διαμορφώνεται εδώ και λίγα χρόνια ε, για την μείωση της παρέμβασης το περιορισμό της παρέμβασης ίσως να ήταν ιδιαίτερα πρόωρο και να οδηγεί σε διακύμανση των τιμών και σε αβεβαιότητα όσον αφορά τους παραγωγούς. Γι' αυτό θα ήθελε οι επιρογνώμονές μας να το σκεφτούν ε, λίγο παραπάνω το θέμα αυτό, να δούμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και η συζήτηση και για το Γάλλο ήταν πολύ σημαντική Είχαμε και τα συμπεράσματα τη υψηλού επίπεδου ομάδα ε, που μα είπαν ότι πρέπει να είμαστε πιο καινοτόμοι για να εξασφαλίσουμε τα εισοδήματα στον τομέα αυτό. Ρωτώ λοιπόν του εμπειρογνώμονε, μήπω πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, του τα συμπεράσματα αυτά σε κάποιου τομεί και σε ποιο βαθμό και αν εσεί αυτή την επέκταση αυτών των μέτρων την στηρίζετε. Τέλο, ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 8, είδαμε πως κάποιοι κερδοσκόποι άλλαξαν ε, το πεδίο δράσης τους από την αγορά αξιογράφων στην αγορά τροφίμων εκμεταλλευόμενοι τις διακοιμάνσεις, αυξάνοντας τις διακοιμάνσεις τελικά, αυξάνοντας την ε, τιμή των πρώτων υλών. Ο Σαρκοζή τελευταία ε, πρότεινε και η συζήτηση γίνεται και σε άλλες χώρες ρύθμιση στο, στη G20 της αγοράς τροφίμων κάτι που γίνεται και στις χρηματοπιστωτικές αγορές αν εσείς έχετε σκεφτεί αυτό το θέμα, αν έχετε κάποιο συμπέρασμα το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει σε σχέση με την πρόταση, η οποία είναι επίκαιρη αυτή την εβδομάδα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ε, Πάρα πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ε, ομιλητών. Θα δώσω επομένω το λόγο τώρα στους επιρογνώμονές μας. Δύο λεπτά. Κατά κεφαλή. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω για μια ακόμη φορά να προσπαθήσω να απαντήσω σε, ένα τα σε κάποια από τα πολλά αριθμά ερωτήματα. Ένα από τα ερωτήματα ήταν κατά πόσο η εμπορική πολιτική θα πρέπει να ενταχθεί στην κοινή γεωργική πολιτική. Στην παρέμβαση μου είπα ότι στην, ε, στη δική μας τη Σαμοσπονδία θεωρούμε ότι όλα διασυνδέονται μεταξύ τους και δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε ξεχωριστά και δεν θα το περιόρισα στην εμπορική αλλά θα συνεπεριλάμβανα την ε, έρευνα, ε, το περιβάλλον ε, και άλλες, την καινοτομία και άλλες πολιτικές. Τώρα, παρατηρήσεις και ερώτηση για τις, τα σούπερ μάρκετ, η διαφάνεια. Θα μπορούσα να σας ανακοινώσω κιόλας ότι εμείς προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε ένα στοιχείο διαφάνεια συζητώντα με τους εταίρους μας ε, στο, κατά μήκο της αλυσίδας και κάναμε και μια έρευνα στα κράτη-μέλη, στα μέλη μας μάλλον, και παρά το πολύ στενόχρονο διάγραμμα είχαμε πάνω από 600 απαντήσεις σε αυτή την έρευνα. Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ε, δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμου. Τους ρωτήσαμε αν ε, υπάρχουν κάποιες αθέμητες εμπορικές πρακτικές που πλήττουν τις επιχειρήσεις αυτές. Ίσως αυτό δώσει μεγαλύτερη διαφάνεια και ίσως και κάποιοι άλλοι στο πλαίσιο της αλυσίδας αυτής θα μπορούσαν να το ελέγξουν. Νομικοί επίσης νομομαθείς θα μπορούσαν να το κοιτάξουν οι ομότιμοι, αλλά εμείς γενικά ως βιομηχανία βρήκαμε κάποιες απαντήσεις και την μελέτη αυτή θα την ε, δημοσιεύσουμε και στην πλατφόρμα Business to Business. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα και το κατά πόσο θα πρέπει και αυτά να ανταποκρίνονται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θέμα δύσκολο. Και πρέπει να σας πω ότι ναι, θέλουμε να είμαστε δίκαιοι φυσικά. Δεν μπορούμε από τη μια πλευρά να περιμένουμε από τους ε, γεωργούς ε, και όλες τους άλλους κλάδους ε, να υπόκεινται σε διάφορους κανονισμούς, κανόνες, πρότυπα. Τα εγκρίνω όλα αυτά, ναι, αλλά αν αυτά δεν τα εφαρμόζουν και οι εκτός της Ένωσης, λυπούμε, αλλά δεν μπορούσατε να περιμένετε τα δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ερώτηση η οποία επανέρχεται από πολλά μέλη του, της Επιτροπής σας η αφορά τις ε, εισαγωγές και τις εμπορικές πρακτικές. Κάποιος αναφέρθηκε στη Μερκοσούρ αλλά και σε, όλα, σε όλες τις εμπορικές πολιτικές. Εγώ σαν Κοζεκά μπορώ να σας απαντήσω σαφέστατα. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να έχουν το κουράγιο να είναι συνετοί ε, σε, για την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση διότι η γεωργία δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει για όλους ό, όπως έγινε τα προηγούμενα 20 χρόνια και ένα σύστημα είναι θα ήταν να πούμε ότι για τα τρόφιμα τα οποία εισάγονται, που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά, περιβαλλοντικά και ίχνης λεσιμότητας με τα ευρωπαϊκά, θα πρέπει μάλλον να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα, με τα εγχώρια θα πρέπει να, είμαστε, θα πρέπει να έχουμε το κουράγιο να είμαστε θαραλέοι, διότι αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τους Ευρωπαίους παραγωγούς μας. Και σε σχέση με τις προβλέψεις που έκανε η ΦΑΟ τα τελευταία, το τελευταίο καιρό, δηλαδή μέχρι το 2050 θα υπάρχει μία διατροφική ανάγκη κατά 70% μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε τώρα θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η διατροφική ανάγκη δεν ε, αφορά μόνο την ποιότητα, δεν θα έχουμε ποσότητα, συγγνώμη, δεν θα χρειαζόμαστε ε, παραπάνω ποσότητα, θα χρειαζόμαστε και ποιοτικά προϊόντα και περισσότερη ποιότητα δηλαδή. Εξού και η δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν φτάσει το, τα υψηλότερα ποιοτικά στάνταρ. Επομένως, ε, θα πρέπει και τα θεσμικά όργανα να σεβαστούν αυτή την ποιότητα. Γι' αυτό η ποιότητα θα πρέπει να μπει στην συζήτηση των ε, ε, θεσμικών οργάνων. Η γεωργία είναι η πηγή, αν θέλετε, όλων των άλλων τομέων. Εξού και θα πρέπει να έχουμε την ε, περηφάνεια να θεωρήσουμε και να επαναφέρουμε την ε, γεωργία πάλι στον πυρήνα και μας το δίνει η, συνθήκη της ε, Λισαβόνας το, αυτή τη δυνατότητα. Βεβαίως, δεδομένων των προβλημάτων με την αστάθεια των τιμών και ε, τα εισοδήματα των γεωργών έχουμε υπερβεί τα όρια με την απελευθέρωση των αγορών και είναι τώρα πολύ δύσκολο να δώσουμε λύσεις σε αυτό το τομέα. Πού θα υπάρξουν λοιπόν αλλαγές. Στο G20 θα συζητηθούν λύσεις θα συζητηθούν και σε άλλες ε, κατευθύνσεις πέραν της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργίας αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να εμπλακεί και η Γεωργία και στα πλαίσια της γεωργικής πολιτικής δεν μπορούμε να δεχθούμε να ε, δίδει κανείς τόσο λίγη σημασία στο θέμα της ρυθμίσεως των ε, μέτρων της αγοράς. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό από τον πρώτο πυλώνα πρέπει να ξαναέρθει στο προσκήνιο και να υπάρξει ένας προπολογισμός ο οποίος από πλευράς ε, διαχειρίσεως αγορών θα καλύψει 2, 3, 4, 5% του προπολογισμού το οποίο δεν επαρκεί για να υπάρχει μια συνεκτική πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια αλλαγή των πολιτικών. Δεν πρέπει κανείς να τις περιλάβει ε, στο δεύτερο πυλώνα όπως της ασφάλειας που δεν έχουν καμία θέση ε, το λέω αυτό παρεπιπτόντος και βεβαίως θα πρέπει να κοιτάξουμε να υπάρξει μία γρήγορη ανταπόκριση από τις δημόσιες αρχές μία βελτίωση της διαφανείας όσον αφορά όλες τις κινήσεις στη διατροφική αλυσίδα. Ε, επίσης όσον αφορά την οργάνωση των γεωργών μπορεί να βοηθήσει αλλά οι γεωργοί ακόμη και οργανωμένοι βρίσκονται απέναντι σε ένα μόνο γαλακτοκομείο, σε ένα μόνο βιομήχανο, οπότε και εκεί θα χρειαστούν τη στήριξη των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Σπάν έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, ε, υπερεύει με τα όρια με την παγκοσμιοποίηση και την απελευθέρωση, όχι γιατί ήταν ελαθασμένες οι απαντήσεις ή γιατί είπαμε όλα είναι ωραία και έτσι θα μείνουν, αλλά διότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις αλλαγές, αλλά υπάρχουν εμπειρογνώμονες και εμείς εμπειρογνώμονες είμαστε, οι οποίοι απαντούν στα γρήγορα, χωρίς προηγουμένως να έχουν παρατηρήσει την πραγματικότητα και εγώ είμαι υπέρ της αποθήκευσης κυρία Γέγκλε ε, και ξέρω ότι ήταν 1,12, 1,6 το μιλήσατε για το γάλα μπορούμε να μιλήσουμε και για το χοιρινό κρέας ε, υπάρχουν διάφορα θέματα που δεν λειτουργούν και υπάρχει μία φούσκα με ε, τις οικοδομές αλλά δεν πρέπει κανείς να λύσει το θέμα χωρίς να υπάρξει εναλλακτική λύση και βλέπουμε ότι εγώ πιστε, πληρώνω για το σιδηρόδρομο για το ειστήριό μου τώρα ένα μεγάλο ποσό σε σχέση με την τιμή του γάλακτος άρα όλα τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν και ο καθένας θα πρέπει να θυμηθεί ποιοι ήταν οι στόχοι μας. Παράγουμε καλά προϊόντα και θέλουμε να συνεχίσουμε να τα παράγουμε. Ε, θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ε, ζωής. Αλλά οι συνθήκες αλλάζουν τόσο πολύ ώστε ε, οι γαλακτοκόμοι έχασαν πέρυσι στο κρατήδιό μου 80% της παραγωγής μας. Αν δούμε την κατάσταση στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία βλέπω ότι υπάρχει μια κατάσταση που επίσης δεν είναι καλή και πρέπει και σε αυτούς κάτι να απαντήσουμε θετικό. Ε, εάν δεν προσπαθούσουμε λοιπόν να αλλάξουμε τα πράγματα με μία μονοκονδυλιά από τη μια μέρα στην άλλη θα πρέπει να προχωρήσουμε και ε, να υπάρξουν ε, μέτρα με, νέα, με νέες δυνατότητες. Διέκοψε τον ομιλητή ο πρόεδρος. Η Μέριεντ ρώτησε γιατί έγινε αυτή η συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Εγώ νομίζω ότι είναι πολιτική. Ε, ε, δόθησαν υποσχέσεις, κρυφά τέλος πάντων η μελέτη αντικτύπου είναι ανεπαρκής, ανεπαρκέστατη θα έλεγα, τι πρέπει να κάνουμε. Την πρωτοβουλία την έχει η νομίζω. Οι διμερείς ε, ε, συμφωνίες είναι αναποτελεσματικές πιστεύω. Έγινε ένα σεμινάριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, αλλά πολύ λίγοι δυστυχώ βουλευτέ πήραν μέρο. Τώρα, η διατροφική αλυσίδα, η διαφάνεια δεν είναι επαρκή. Ε, η αλυσίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολλοί άνθρωποι τρώνε από αυτήν. Οι πολιτικές ανταγωνισμού πιστεύω ότι δεν είναι προσαρμοσμένες ε, έτσι ώστε να βελτιώσουν την ε, κατάσταση. Η διακύμανση, οι αγορές των προϊόντων κατανάλωσης συνδέονται όλο ένα και περισσότερο με τις ε, οικονομικές αγορές, οι οποίες ε, παρουσιάζουν μια μεγάλη, είναι πολύ ευμετάβλητες. Επίσης ε, για τα, ποιοτικά, για τα ποιατικά πρότυπα και το, το περιβάλλον. Τα επιβάλλουμε στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να, να, το, να τα εφαρμόσουμε και στις άλλες, σε άλλες χώρες. Εάν δεν υπάρχει όμως αμοιβαιότητα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ε, με την Μερκοσόρ, τι λέμε, θα, λέμε θα εισάγουμε περισσότερα γεωργικά προϊόντα και ξέρουμε ότι το περιβάλλον ε, στις χώρες σας θα καταστραφεί, θα ε, εξαφανιστεί το τροπικό δάσος. Αλλά μην ανησυχείτε, θα το προσέξουμε. Ε, γλυφιτζούρια τέλο πάντων όλα αυτά. Τώρα όσον αφορά την διαχείριση των τον του κινδύνου. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν καλές προτάσεις εδώ. Ευχαριστώ Κοράντο. Ο κύριος Ντόουερ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι κάποιος είπε ότι πρέπει να δούμε και τους άλλους εμπλεκομένους στη διατροφική αλυσίδα. Και η CIA κοιτάζει και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις συμβατικές σχέσεις και στους όρους πληρωμής προς τους προμηθευτές. Υπάρχει μια γενική αρχή εδώ η οποία δεν έχει αναφερθεί που είναι η σπατάλη σε τρόφιμα διότι ένα τρίτο των τροφίμων παράγοντα στην Ευρώπη πετιούνται. Λοιπόν, πρέπει να ελέγξουμε πού συμβαίνει αυτό στη διατροφική αλυσίδα και συνήθως είναι οι εμπορικές μέθοδοι στη διατροφική αγορά. Όσον αφορά τον καταναλωτή, αυτά τα οποία λέμε στις διαβουλεύσεις που ξεκίνησε ο Επίτροπος όλος, όταν μας λέγουν ότι ενδιαφέρονται για την ποιότητα των τροφίμων, το περιβάλλον, ότι το εισόδημα των γεωργών όλα αυτά εκφράζονται στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αγοράζουν τρόφιμα. Όταν λοιπόν γνωρίζουν ποιες είναι οι προδιαγραφές των ευρωπαϊκών τροφίμων και των αλλοδαπών πόσο ποσοστό από την τελική τιμή ε, πληρώνεται στους γεωργούς από το σύνολο που κοστίζει στο κατάστημα ίσως θα αγόραζαν κατά τρόπον ώστε να πρημοδοτήσουν τους γεωργούς. Επίσης ε, αναφέρομαι και στις δημόσιες αγορές ε, για τις τοπικές, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τις κυβερνήσεις οι οποίοι μπορούν να αγοράσουν κατευθείαν από τους γεωργούς με καλή ποιότητα. Δεν χρειάζεται να αγοράζουν ότι είναι φτηνότερο για να δώσουν το καλό παράδειγμα καλή συμπεριφορά στην διατροφική αλυσίδα. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα, ευχαριστώ όλους ε, και περνάμε στην τρίτη συνεδρία στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Τρεις ερωτήσεις και θα ζητήσω, θα διαβάσω τις τρεις, τρεις ερωτήσεις και θα ε, απαντήσετε κι εσείς με τη σειρά σας. Πρώτη ερώτηση. Θα αντικατασταθεί ο κύριος με τον πρόεδρο της ε, Κοζέκα με τον πρόεδρο της ε, κόπα. Ο κύριος Μπρούνι θα αντικατασταθεί με τον κύριο Walsh. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση, πώς θα πρέπει οι, στόχοι αξιολόγηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνική και οι, εφαρμο... προτεραιότητες εφαρμογής να οριστούν γιατί και τα μελλοντικά προγράμματα ανάπτυξης της Υπέθρου. Ε, δεύτερη ερώτηση, συμφωνείτε με την ε, προσέγγιση της ε, Επιτροπής για τις, όσον αφορά τις πληρωμές και την υποστήριξη ε, για συγκε, με, λαμβάνοντας υπόψη ε, τις συγκεκριμένες, ε, τους συγκεκριμένους φυσικούς περιορισμούς και πώς θα πρέπει να ενισχυθεί η ενίσχυση ανάμεσα στην ανάπτυξη της υπαίθρου και τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Ο κύριος Walsh. Οι, οι περιοχές της υπαίθρου καλύπτουν πάνω από το 1 τέταρτο της ευρωπαϊκής επικράτειας και υπάρχουν μεγάλες διαφορές και πολύ σημαντικές μάλλον οι περιοχές αυτές ε, για την ε, ανάπτυξη της ε, Ευρώπης, όμως παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. Άλλες είναι εύρωστες, άλλες έχουν, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Οι περιοχές αυτές έχουν υλικό, αν θέλετε, και ανθρώπινο και φυσικό ε, υλικό, το οποίο είναι πολύτιμο για, την, ε, για το μέλλον της Ευρώπης. Επομένως, θα πρέπει να, ε, το, να ενισχύσουμε την Επιτροπή, την ανάπτυξη της επίτησης Πέτρου. Θα πρέπει να ορίσουμε στόχους για νέα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και θα, η απάντηση είναι για μας ο, ο, ο συσχετισμός όλων των ταμείων ε, ε, με την ε, ανάπτυξη της Υπέθρου. Οι διάφοροι επίτροποι, τρεις επίτροποι βασικά, μεταξύ αυτών και η κυρία Δαμανάκη, έγραψαν μια επιστολή στον κύριο Μπαρόσο για το νέο στρατηγικό πλαίσιο για αυτά τα πέντε διαρθρωτικά ταμεία. Εμείς υποστηρίζουμε αυτή την προσέγγιση. Εάν θέλουμε να δράσουμε σε, τρία επίπεδα, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό, θα πρέπει να ε, απλουστεύσουμε τις διαδικασίες, γι' αυτό ζητάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει μια, ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τα πέντε ταμεία τα οποία ανέφερα, οι κανονισμοί για αυτά τα, νέα, για αυτά τα πέντε ταμεία πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένοι μεταξύ τους και ε, θα πρέπει να υπάρχει μια απέτηση τα εθνικά και τα περιφερειακά ε, και να έχουν τα δικά τους ε, πλαίσια τα οποία να αντικατοπτρίζουν το κοινοτικό πλαίσιο και στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, και Αλίας ε, θα πρέπει να ε, υπάρχουν περαιτέρω χρηματοδοτήσεις, περαιτέρω κονδύλια για μια συνεργασία ανάμεσα στους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς έτσι ώστε να υπάρχει στρατηγική ανάπτυξη της υπαίθρου χρησιμοποιώντας όλα τα εθνικά ή ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτό βέβαια θα ξεπεράσει, πιστεύουμε, και την, ε, τα επιτυχημένα προγράμματα Leader. Επίσης θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη, η καινοτομία, τεχνολογία που θα οδηγήσει σε μια αναγέννηση της υπαίθρου και της γεωργίας. Ευχαριστώ. Τον λόγο τον έχει ο Κοράντο Πίτσιο Μπίρολη Θα είμαι πιο σύντομος, δύσκολο για να είναι αλλά τέλος πάντων. Πώ θα πρέπει οι στόχοι αξιολόγηση εθνική και κοινοτική να ορίζονται. Οι υφιστάμενε διαδικασίε και δομέ είναι αχρίαστα πολύπλοκες για του ε, υπεύθυνου διαχείριση και πολλέ από τι διαδικασίε ε, υποβολή αιτήσεων είναι πάρα πολύ δύσκολε και για του ίδιου του ετούντε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν προσπάθειε απλούστευση στον τομέα αυτό. Αναγνωρίζουμε επίση ότι τα μέτρα τη κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να έχουν ε, σαφούς, σαφείς στόχους και να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησής τους και αξιολόγησης της επίτευξης και του, της καλύτερης δυνατής ε, εφαρμογής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την ε, top-down προσέγγιση, δεν ήταν πολύ υπέρ Ευρωπαϊκή Ένωση για το πλαισιο 2015 2007-2013. Υποστηρίζουμε να αλλάξει η προσέγγιση. Δηλαδή, να συμφωνηθούν στρατηγικοί στόχοι σε κοινοτικό επίπεδο και μετά τα κράτη-μέλη να κληθούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προσαρμόσουν στις δικές τους ιδιαιτερότητες και βέβαια επιτόπου μετά οι αγρότες να δουν πώς πιο αποδοτικά και με το μικρότερο κόστος μπορούν να εκμεταλλευτούν και τις τοπικές τους ε, γνώσεις. Πρέπει σε όλα αυτά να έχουμε υπόψη μας ότι τα εθελοντικά μέτρα μπορεί να μην εφαρμοστούν εάν οι αγρότες δεν θεωρήσουν ότι υπάρχει ε, θετική κόστου κόστους-οφέλους. Και ό,τι και αν λέμε και κάνουμε στην αγροτική ανάπτυξη δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα αν δεν έχει αυτό όφελος για τους ίδιους τους αγρότες. Δεν θα το κάνουν ποτέ. Δεν μπορούμε να προβλέπουμε κανονισμούς και να λέμε ορίστε υπάρχει κανονισμός και πρέπει να τον ακολουθήσετε γιατί αυτό συνεπάγεται κόστος. Το ερώτημα λοιπόν είναι μπορεί, θα εφαρμοστεί ή όχι ο κανονισμός. Πρέπει το, τη ρύθμιση τους κανονισμούς να τους συνδυάζουμε με κίνητρα αυτό είναι σημαντικό για τους αγρότες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κοράντο. Σαβινή τώρα. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ασχοληθώ με το τρίτο ερώτημα συνεργασία δηλαδή μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Και εμείς νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια συνέπεια στους διάφορους στόχους και αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο περιοχών για να υπάρχει συνεργασία και καλή αποτελεσματικότητα στο επίπεδο των ταμείων. Φαίνεται σημαντικό επίσης να υπάρχει μια προσέγγιση εδαφική, δηλαδή οι διάφοροι φορείς να μπορούν να συζητούν τα βασικά διακυβεύματα, δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση, διάφορα επίπεδα κυβέρνησης, γεωργοί αγρότες, αλλά και οι άλλοι φορείς που ασχολούνται παραδείγματος χάρη με το περιβάλλον, ώστε να υπάρχει μια συντονισμένη δράση που όλοι θα την καταλαβαίνουν και θα ανταποκρίνεται καλά τα όσα διακυβεύονται. Τώρα, τι διακυβεύεται για μας, το ξαναείπαμε όταν τοποθετήκαμε πιο γενικά πιο ε, εντοπισμένη, αν θέλετε, γεωργία, πιο κοντά στον πολίτη, ποιοτική γεωργία που να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις προκλήσεις του σήμερα. Άρα, για να ευνοήσουμε την ποιότητα, καλό νομίζω είναι να έχουμε προσέγγιση και κατάρτισης και καινοτομίας και έρευνας πιο οικολογικών τρόπων παραγωγής. Σημαντικό είναι επίσης να δούμε το θέμα της ποιότητας, σχέση ποιότητα τροφίμων και υγεία. Σε μια εδαφική προσέγγιση μπορούμε να δώσουμε καλύτερη απάντηση ε, στις ανάγκες των διαφόρων φορέων, σχολεία, λύκεια. Όσοι μέσω της συλλογική διατροφής ε, μπορούν να επηρεάσουν και την υγεία των ανθρώπων που θα καταναλώσουν τα τρόφιμα αλλά και τους αγρότες που θα μπορούν να προσαρμόζουν την παραγωγή τους στις τοπικές αγορές. Και σε ό,τι αφορά τα διακυβεύματα θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη διασύνδεση αστικών κέντρων και υπαίθρου για να μην υπάρχει αυτό το χάσμα ε, που υπάρχει μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου. Οι πόλεις όλο και δυσκολότερα καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στην υπαίθρο και αυτό επηρεάζει την καλύτερη κατανόηση της διτροφικής αλυσίδας. Τι γίνεται τι επίπεδο έχουν οι τιμές και τα λοιπά. Αυτή η πολιτική προσέγγιση εγκύτητας σε ορισμένες χώρες μπορεί να βοηθήσει να επανακατακτηθούν κάποιες αγορές 50 έως και 60% των προϊόντων που μπορεί να βρει κανείς στα σούπερ μάρκετ εισάγονται σε ορισμένες χώρες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό στους τοπικούς παραγωγούς λοιπόν είναι σημαντική πρόσβαση στην τοπική αγορά αλλά και μέσα από κλασικές αλυσίδες που θα είναι όμως προσαρμοσμένες στους παραγωγούς των περιοχών αυτών. Αυτά είναι τα βασικά. Αυτό που θεωρούμε πολύ σημαντικό πάντως είναι η μελλοντική ΚΑΠ να είναι προσαρμοσμένη και στους παραγωγούς αλλά και στους καταναλωτές, στους πολίτες. Γουόλς τώρα, κόπα, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες μας ε, υποστηρίζουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για αυτές ε, τις κατευθυντήριες γραμμές, αυτά τα θέματα, καινοτομία, κλιματική αλλαγή και βέβαια περιβάλλον, αλλά θέλουμε να προσθεθεί και ένα τέταρτο θέμα, πρόθεση ανταγωνιστικών, αποδοτικών ε, εκμεταλλεύσεων και αγορο... ενώσεων παραγών. Ίσως δεν υπάρχουν ούτε και δύο εκμεταλλεύσεις που να έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες μπορεί κάποια πτυχή που θεωρείται σημαντική σε μια περιφέρεια να μην θεωρείται σημαντική σε μια άλλη. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητε. Και αυτή είναι μια καλύτερη προσέγγιση και όχι να εφαρμόζονται ομοιόμορφα τα πάντα. Τώρα, θέλουμε να βασιστούμε στην έκβαση, στο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να μπορεί να υπάρχει και μια σωστή μέτρηση των αποτελεσμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση σε όλες τις περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τι πληρωμές τώρα στις λιγότερο ευνεμένες περιοχέ, νομίζουμε ότι πρέπει αυτό να παραμείνει στο δεύτερο πυλόν. Και μας ανησυχεί η νέα οριοθέτηση αυτών των περιοχών από την Κομισιόν. Και επειδή υπάρχει και πληρωμή επιπλέον στο πλαίσιο του πυλώνα 1, θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου. Γιατί αν ισχύσει ομοιόμορφα θα φτάσουμε στα 10 ευρώ ένα εκτάριο, κάτι που δεν έχει καμία σημασία δηλαδή για τους αγρότες. Νομίζουμε επίση ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη συνέπεια μεταξύ των μέτρων της κοινή γεωργική πολιτικής για την ανάπτυξη τη Πέδρου και άλλων μέτρων που μπορεί να έχουν εδαφικό αντίκτυπο. Η κοινή γεωργική πολιτική πιστεύουμε είναι αρμόδια για τη γεωργία. Πρέπει να εξασφαλίσει την συνεκτικότητα, τη συνέπεια μεταξύ περιοχών. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας για τη συμμετοχή της γεωργίας αλλά και της δασοκομείας βέβαια στην ανάπτυξη της ΥΠΕΔ. Χαιρετίζουμε την έμφαση που δίνεται στην έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό για τη γεωργία αυτό λόγω των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ιδίω γιατί έρευνα και καινοτομία είναι ο καλύτερο τρόπο να βοηθήσουμε του αγρότε να ανταποκριθούν ε, στι ανάγκε και να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει και στον τομέα του περιβάλλοντο και σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματο και βέβαια θα πρέπει να παραμείνουμε και ανταγωνιστικοί. Μα ενθαρρύνει η δέσμευση του Επιτρόπου για τα ερευνητικά προγράμματα που λέει ότι θα αναλάβουν αυτή την πρόκληση. Ο ρόλο τη ΚΑΠ πρέπει να είναι να εξασφαλίσει όχι μόνο να γίνεται η έρευνα, αλλά και να έχει αποτελέσματα επιτόπου στι γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Και βέβαια θα πρέπει να κεντρωθούμε στην πολλαπλή συμμόρφωση. Ολοκληρώνοντα, θέλω να πω ότι αν στην Ήπεθρο δεν ζουν και δεν εργάζονται και δεν κερδίζουν χρήματα... Έκλεισα το μικρόφωνο. Σπάν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς είμαστε υπέρ μιας πολιτικής δύο πυλώνων ε, και μια ανεξάρτητη αυτόνομη ανάπτυξη του χώρου της υπέδρους. Χρειάζονται και άλλες πολιτικές ε, διότι προς το παρόν βασίζεται κανείς ε, στην πολιτική για τις, μεγάλες πόλεις και δεν ασχολείται επαρκώς με την Ήπεθρο. Εάν λοιπόν η διαρθρωτική πολιτική και η περιφερειακή πολιτική αυξηθούν από πλευράς αριθμών τότε θα υποφέρει η Ήπεθρος και η γεωργική πολιτική και ουσιαστικά η παραγωγικότητα της Ήπεθρου είναι μεγαλύτερη από τον πόλο και γι' αυτό ζητούμε να υπάρξουν εγκαίρως διάφορες διασυνδύσεις μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τρόπον ώστε να συνδυαστούν οι προσπάθειες και να μπορέσει ε, ο συλλογικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλλει σε μία ε, μεγάλη ε, σε ένα μεγάλο οικοδόμημα ευρωπαϊκών μέτρων για να μπορέσει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε αντίθετοι εν πάση περιπτώσει σε αυτό το οποίο προτείνεται εδώ. Και ε, όσον αφορά το θέμα της ε, έρευνας, ε, σωστά ελέγχθη ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα και θα πρέπει να αξιολογήσουμε και τα αποτελέσματα των μέτρων τα οποία εφαρμόζονται στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη μεγαλύτερη δικτύωση διότι η Ευρώπη είναι πολύ επιτυχή στην Ήπεθρο και για την έρευνα υπάρχουν πολλά ενάψματα για να μπορέσει κανείς να προωθήσει τα αποτελέσματα από ένα χωριό προς τα έξω αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει τα εγχειρήματα αυτά και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα και κάτι πρέπει να είναι σαφές ότι η γεωργία θα πρέπει να προωθηθεί στον πρώτο πυλώνα για να δούμε με τι βάσεις και τι κριτήρια και ποιους δείκτες θα προχωρήσουμε αλλά χρειαζόμαστε τον δεύτερο πυλώνα στη γεωργία και εντός και εκτός της γεωργίας ε, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και τις άλλες πολιτικές για να τις στηρίξουμε. Ε, επίσης ε, η εκπαίδευση πρέπει να παραμείνει στο δεύτερο πυλώνι και να ενισχυθεί. Σας ευχαριστώ. Και τώρα... Ερχόμαστε στο τελευταίο τμήμα των παρεμβάσεων. Ευχαριστώ όλους. Βλέπω ότι έχουμε 7 εγγεγραμμένους στον κατάλογό μου. Δύο λεπτά ο καθένας. Με συγχωρείτε. Ξέχασα την κυρία Φρέιουελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Αφενός, οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν ενδιαφέροντα μέτρα για αύξηση της αγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Θα πρέπει να δυναμωθούν τα μέτρα αυτά. Συμφωνούμε. Αφετέρου όμως η επέκταση των μέτρων που το τα κράτη-μέλη θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει σε επανακρατικοποίηση. Και όπω είπα, εμεί δεν είμαστε υπέρ αυτή τη προσέγγιση. Η διατήρηση μια ενίας αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα πρέπει να είναι ο γνώμονα που θα διέπει τη μελλοντική ΚΑΠ. Ο δεύτερο τώρα πυλώνας περιλαμβάνει επίση πολύτιμα μέτρα για την αύξηση τη ανταγωνιστικότητα τη αγροδιατροφική αλυσίδα ή επενδύσεις σε νέες τεχνολογίε, εξυγχρονισμό, μέτρα για την πρόθεση της γνώσης, τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, ενθάρρυνση συμμετοχή των αγροτών σε ποιοτικά συστήματα, σε συστήματα ποιότητα, όλα αυτά είναι καλά μέτρα και θα έχουν αποτέλεσμα. Επίσης, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το ότι η φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση της ε, αγροτικής πολιτικής είναι να γίνει μέσω μιας στοχευμένη πολιτική και στοχεύει στα αποτελέσματα, στην έκβαση και όχι στον τρόπο. Και αυτό είναι πολύ καλό σε ό,τι αφορά την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ ανάπτυξης Πέθρου και των άλλων πολιτικών. Το έχω προαναφέρει. Ο Επίτροπος Τσιόλος είπε ότι συνεργάζεται με άλλους επιτρόπους ε, για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ΚΑΠ και πολιτικής έρευνας. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ίσως πρέπει να πάει και ένα βήμα παραπέρα, να μιλήσει και με άλλους επιτρόπους, όπως είναι ο Επιτρόπος Ντάλι ή ο Επιτρόπος Ντεχούχτα και το περιβάλλον, τον αρμόδιο επίτροπο και ενέργεια, βιοκαύσιμα. Δεν το ακούσαμε και πολύ να αναφέρεται το θέμα αυτό σήμερα. Αλλά νομίζω ότι στόχος βασικός της πολιτικής της γεωργικής είναι η παραγωγή πρώτων υλών για τρόφιμα και ζωοτροφές στην Ευρώπη. Και η γεωργική πολιτική έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο υπέρ της καινοτομίας, μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ ΚΑΠ και ερευνητική πολιτικής και είναι μια καλή κατεύθυνση αυτή. Και μπορώ εδώ να σταματήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μέλα και ζητώ συγγνώμη κιόλα. τελειώνουμε με, τον, με, τους, με τα μέλη της Επιτροπής μας, ο η κυρία Πόλσεν αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε όταν μιλάμε για περιοχές της υπαίθρου, προφανώς χρειάζεται μία βοήθεια. Βοήθεια όμως για τις επενδύσεις κυρίως. Και πιστεύω ότι μία συνεργασία ανάμεσα στα ταμεία, στα διαρθρωτικά ταμεία, στο, στο Ταμείο Συνοχής και τον δεύτερο πυλώνα είναι απαραίτητη. Κυρίως όσον αφορά το capital risk. που αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου και την γεωργία. Εγώ ζω σε μια περιοχή που είναι μεγαλύτερη από το Λουξεμβούργο με 10.000 κατοίκους όπου ε, το κοντύτερο, το πιο κοντινό γαλακτοκομείο είναι 250 μέτρα. Δεν μπορούσα να θεωρώ, δεν, νομίζω ότι είναι λιγότερο ευνοημένη περιοχή αυτή, κυρίως να μιλάμε για μικρές εκμεταλλεύσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν μικρές αγορές, τοπικές αγορές, αγορές που να έχουν μία υποδομή. Δεν θέλουμε να, δημι... να να ενισχυθούν οι εκμεταλλεύσεις. Απλώς αυτό το οποίο θέλουμε είναι η κάθε εκμετάλλευση να έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Η Ελίζα Μπεθ Κόστιγκερ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι Αυστριακή, μια χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από την ε, δομή των μικρών αγροκτημάτων και υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν λεφθεί ιδίως για τις μειονεκτικές περιοχές και για τις ορεινές περιοχές. Ε, υπάρχει, θέλουμε, έχουμε σαν στόχο να αυξήσουμε και κατά 30% το ποσοστό των βιολογικών καλλιεργειών. Ε, θα πρέπει λοιπόν ορισμένες περιοχές ε, που έχουν ειδικές, ειδικά χαρακτηριστικά να αναγνωρίζονται στα πλαίσια της επικουρικότητος. Πώς εσείς αξιολογείτε το screening της πρώτης, του πρώτου πυλώνα σε αυτό το τομέα και πώς ε, πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της γύρανσης στον τομέα της γεωργίας και πώς να το επιλύσει. Επίσης τι γίνεται με κράτη ε, τα οποία απορρίπτουν ε, την συγχρηματοδότηση και την χρήση του δευτέρου πυλώνα. Πώς είναι δυνατόν όλες οι χώρες να έχουν τη σωστή πρόσβαση στα μέτρα Τη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ε, κατ' εμέ πρέπει να υπάρχει στήριξη της γεωργίας αλλά να κρατηθεί ε, ζωντανή και η ύπερθρος, οπότε πιστεύω ότι τα κρατικά μέτρα πρέπει να καταδικαστούν. Ο κύριος Ταμπατζή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να πω, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης υπέθρου, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εναρμόνισης ανάμεσα στις γεωργικές πολιτικές και στις αναπτυξιακές πολιτικές. Στην, όταν μπήκε η Ουγγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η, η Ουγγαρία είδαμε ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου ήταν ένα σημαντικός τομέας της πολιτικής. Όμως, πολύ σημαντική, είναι πολύ μεγάλη η, ε, η ανεργία στον, στον τομέα, στην περιοχή αυτή. Ε, προβλήματα με, τις, με το δικό δίκτυο, ε, με τη διαχείριση των υδάτων. Σε αυτό σε όλες τις χώρες που προσχώρησαν τότε εκείνη την περιοχή. Ε, επομένως, τα επόμενα, τα επόμενα χρόνια, μετά το 2014, θα πρέπει να ισχύσει, θα ισχύσει μάλλον και θα, και θα, είναι, θα είναι υποχρεωτικό να έχουμε μια διαφοροποιημένη ε, γεωργική πολιτική η οποία να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές ε, ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη και θα είναι μια πολιτική η οποία θα εισάγει, εισάγει συστάματα, συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον και φιλικά προς το έδαφος θα επιβάλλει την ε, εισαγωγή συγκεκριμένων μηχανημάτων, συγκεκριμένων ε, φυτών Επομένως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη όταν μιλάμε για ανάπτυξη της υπαίθρου, διότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Πορτογαλία και η Ουγγαρία ή και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ και πάλι είναι κρίμα ότι μιλάμε λιγότερο για τον δεύτερο πυλώνα και περισσότερο για τον πρώτο και κατά τη γνώμη μου μπορούμε να διαμορφώσουμε μεγαλύτερες πολιτικές επεμβάσεις από το δεύτερο πυλώνα αλλά η πρόθεση της ανταγωνιστικότητας της Γεωργίας είναι ένα σημαντικό θέμα. Υπήρξε ε, μία εκ των άνω κατεύθυνση η οποία μείωσε τις θέσεις εργασίας, δεν προώθησε και ίσως και κατέστρεψε τις μικρές δομές και πιστεύω ότι εδώ πρέπει να δούμε ε, πώς θα χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο πυλόν με ε, τη δημιουργία λυσίδων οικονομικής αξιοποίησεως ίσως θα πρέπει εδώ να ασχοληθούμε και με το θέμα του εργατικού δυναμικού και το πώς θα, χρησιμοποιήσουμε τους δημόσιους πόρους διότι η δομή με τους πυλώνες ως έχει ε, παραμείνει έτσι αν θέλουμε να πρασινίσει ο πρώτος πυλώνας τότε θα αναρωτηθούμε τι θα γίνει με τον δεύτερο πυλώνα δηλαδή πώς εκεί θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα και το ερώτημα τίθεται ε, αν ε, δεν πρέπει να έχουμε μεγαλύτερες επεμβάσεις ε, σαν πρώτο θέμα διότι ε, πρέπει να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα στον χώρο της υπαίθρου και το τρίτο ερώτημά μου που ήδη έχει τεθεί είναι η συγχρηματοδότηση. Δεν είναι δυνατόν διάφορα προγράμματα που είναι καλά και χρήσιμα για μερικά κράτη να μην προωθούνται λόγω ελλείψεως συγχρηματοδότησης οπότε πρέπει να αλλάζουμε κατά τη ε, ε, εξαρτωμένη της σημασίας ε, τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η συγχρηματοδότηση για να μπορούν να συμμετέχουν όλο και περισσότερα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριε Χόισλινγκ. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Ράιμερς η οικονομική χρήση ε, άφησε ε, τα χνάρια της παντού και επηρέασε τη λήψη αποφάσεων άρα δεν εξαιρέθηκε και η κατάσταση της γεωργίας. Η συγχρηματοδότηση του δεύτερου πυλώνα ε, μπορεί να αποκλείσει την συμμετοχή επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε διαφορετικά τη συγχρηματοδότηση. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο διότι διαφορετικά κλείνουμε το μικρόφωνο και τώρα δίνω το λόγο στον Μίκαελ Βόιτσεκ και με συγχωρείτε αλλά δεν μπορώ να προφέρω το επίθετό του. Ευχαριστώ. Μιλάμε για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό το πρόγραμμα, κατά κύριο λόγο, συνεισφέρει στις συγκέντρωση της παραγωγής σε τεχνολογικές αλλαγές και στην υιοθέτηση τεχνολογιών αχμής σε άμεσα συνδόμε με την παραγωγή περιοχές. Αλλά υπάρχουν και δαπάνες που έχουν να κάνουν με τη μεταποίηση. Τι σημαίνουν όλα αυτά για σήμερα. Σημαίνει μάλλον ότι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ε, τουλάχιστον στην Πολυρία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, μάλλον θα οδηγήσει σε λιγότερες ε, παραγωγικές μονάδες από ό,τι μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ορίσουμε τι στόχο θέλουμε να πετύχουμε. Γιατί από τη μια σήμερα παραπονιέστε ότι υπάρχουν λιγότεροι αγρότες, λιγότερες θέσεις εργασίας, από την άλλη κάθε ευρώ το οποίο δαπανάτε από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για κάθε δράση και για τα περιβαλλοντικά μέτρα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι θέσει εργασία στον τομέα της γεωργίας. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν μπορεί να υπολογιστεί σε κανένα μέτρο, σε καμία δράση. Ακόμη και αν, για παράδειγμα, επενδύσουμε σε δεντροφύτευση παραδείγματος ε, χάρη, οπότε αποκλείουμε ένα μέρος ε, των εδαφών από την καλλιέργεια προϊόντων. Επίση, αναποθέτω πολλέ ελπίδε σε αυτά που ακούσαμε σήμερα, ότι δηλαδή θα πρέπει το πρόγραμμα αγροτική ανάπτυξη να συμβάλλει περισσότερο στην έρευνα και στην εισαγωγή τεχνολογιών εχμή. Επίση, τα προγράμματα αγροτική ανάπτυξη μεταφράζονται στη στήριξη διαφόρων κοινωνικών μέτρων και εκπαιδευτικών εκστρατιών. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχουν περιθώρια λιγμών. Πάντα υπάρχουν περιθώρια λιγμών. Τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόντουστ. Ε, υπάρχουν ε, στενές ε, διασυνδέσεις ε, μεταξύ γεωργίας και υπαίθρου και γι' αυτό χρειάζεται μία ολοκληρωμένη πολιτική για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η δημογραφική εξέλιξη, τα προβλήματα τα κλιματολογικά και τα οι οικονομικές επιπτώσεις. Θα πρέπει ε, να εξετάσει κανείς τις επιχειρήσεις πώς θα οργανωθεί η εκπαίδευση για τους γεωργούς και πώς θα προσελκύσετε κόσμο στην Ήπεθρο διότι εδώ μιλάμε για ε, τους ε, δημόσιους πόρους και για τους στόχους μιλάμε για την ποικιλομορφία θα ήθελα να ξέρω τι θέση θα έχουν τα θέματα αυτά η συγκοινή γεωργική πολιτική και πώς θα χρηματοδοτηθούν από τον πρώτο ή από τον δεύτερο πυλώνα. Και τρίτον, εάν θέλετε να είναι ισχυρή η ύπεθρος, εάν θέλετε η ύπεθρος να μην είναι ένα παραμάγαζο της ε, περιφερειακής πολιτικής είσαστε έτοιμοι να μεταφέρετε πόρους και χρήματα από τον πρώτο πυλώνα στο δεύτερο πυλώνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους. Πριν ε, δώσω το λόγο ε, την, τον λόγο του τέλους στον Άλμπερτ Ντες να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες εάν και εφόσον θέλουν δεν είστε υποχρεωμένοι να πάρετε το λόγο αν θέλετε όμως μπορείτε να παρέμβετε για ένα λεπτό θέλετε να πάρετε το λόγο ο κύριος Walsh για ένα λεπτό Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανάπτυξη της υπαίθρου ήθελα να πω ότι εάν οι παραγωγοί γεωργοί δεν είναι εκεί στην υπαίθρο να, ε, να δουλεύουν και να παράγουν κανείς δεν θα μπορεί να πάρει τα χρήματα από τον δεύτερο πυλώνα. Επίσης, ε, αν θέλουμε να μπουν και νέοι στο επάγγελμα, που είναι, σίγου, που είναι απαραίτητο, ε, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι νέοι θα δουν και ένα μέλλον στην γεωργία. Δηλαδή, θα ε, είναι σε θέση να ζήσουν, να θρέψουν την οικογένειά τους. Αυτό είναι ουσιαστική σημασία. Θα πρέπει να έχουμε έναν ισχυρό πρώτο πυλώνα, όμως θα πρέπει να εργαστούμε και μέσα στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα γιατί εάν δεν έχουν κέρδος ε, από την εργασία και από την διαβίωση στον, ε, ε, στην, Ήπεθρο, τότε θα οδηγηθούμε σε μια απερίμωση της, της Ήπεθρου. να πρέπει να αφήσουμε τους πυλώνες δηλαδή ως έχουν. Ο, Κορά, ο δόκτωρ Κοράντο Πίτσιο Μπίρολη. Η Κομισιόν θα πρέπει να επανέλθει ίσως σε προηγούμενες ε, προτάσεις της, διότι τώρα αυτό το οποίο προτείνει είναι ιδιαίτερα περίπλοκο σύστημα. Επίσης ε, για τις αναπτύξεις ε, περιοχές της υπαίθρου που είναι λιγότερο ευνοημένες δεν θα πρέπει να τις ονομάζουμε έτσι θα πρέπει να τις βρούμε, βρούμε μια άλλη ονομασία πιο θετική Στη συγχρηματοδότηση τώρα θα πρέπει να την εφαρμόσουμε με έναν ευέλικτο τρόπο, διότι αλλιώ θα χάσουμε την Ανατολική Ευρώπη και αν χάσουμε την Ανατολική Ευρώπη θα χάσουμε την δεύτερο πυλώνα. Επομένω κάτι πρέπει να κάνουμε εκεί. Τώρα, στην, στις, στα έργα υποδομή τα οποία δεν υπάρχουν. Είναι το Περιφερειακό Ταμείο εδώ και για τους δύο πυλώνες ε, θα τους χρειαζόμαστε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη, μετα... τη μεταρρύθμιση. Και για την έρευνα χρειαζόμαστε τεχνολογική έρευνα. Δεν, μιλάμε μόνο, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για τα βιοκαύσιμα, ε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαβίνια έχει, έχει το λόγο. Επανέρχομαι στο θέμα των, ε, της καταρτήσεως ζωνών και των ε, μειονεκτικών ζωνών. Εάν ε, δεν υπάρχει σωστή χρηματοδότηση, το θέμα είναι ανησυχητικό. Δεν πρέπει να μειώσουμε τις ζώνες, αλλά να διευρύνουμε τις μειονεκτικές ζώνες. Όσον αφορά τον διαχωρισμό σε δύο πυλώνες, είναι κάπως τεχνητός, αλλά τον καταλαβαίνουν οι γεωργοί και δεν πρέπει να υπάρχει αντίφαξη μεταξύ των στόχων του πρώτου πυλώνα και του δεύτερου. Δεν μπορούμε στο δεύτερο να καταστρέφουμε τους γεωργούς και με το δεύτερο να τους επιτρέπουμε να εγκατασταθούν. Πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα στους στόχους και συμφωνούμε με την ιδέα ότι πρέπει να διατηρήσουμε έναν παρική ε, πληθυσμό γεωργικό για να μπορέσουμε να επεξέλθουμε στις προκλήσεις που υπάρχουν υπάρχουν σήμερα. Ευχαριστώ. Ντάουερ, δύο πράγματα πρέπει να πω. Μου άρεσε που η Αντιπρόεδρος μίλησε για περιφερειακές ε, και τοπικές αγορές. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο μια νέα κοινή αγορά, αλλά και πολλαπλές τοπικές και περιφερειακές αγορές. Καμία δεν είναι απόλυτο στεγανή, στεγανοποιημένη, αλλά Εκεί γίνεται μεγάλο μέρος του τοπικού εμπορίου, των τοπικών συναλλαγών και αυτό ε, έχει μεγάλη δύναμη ε, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Κάτι άλλο. Για το πρόγραμμα Leader είπε κάποιο ότι θα ήθελε να ακούσει περισσότερα. Εγώ έδωσα έμφαση στι λεγόμενε υποπεριφερειακές εταιρικέ σχέσει που νομίζω ότι θα είναι η επικαιροποιημένη έκδοση του Λίντερ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω έχει λόγους να είναι πάρα πολύ υπερήφανη για την πρωτοβουλία Λίντερ και τα αποτελέσματά τη. Ωστόσο, από πολλές πτυχές δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρω. Θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη λοιπόν, να προσελκύσει περισσότερα κονδύλια και να την εμπιστεύονται περισσότερο οι κυβερνήσεις και να έχει και ένα μεγαλύτερο ρόλο όπου μπορεί να τον έχει. Ευχαριστώ. Η Μέλα, ευχαριστώ πολύ, πολύ γρήγορα. Για τους δύο πυλώνες, εμείς στη βιομηχανία των τροφίμων ε, υποστηρίζουμε την διατήρηση και των δύο πυλώνων, γιατί και οι δύο έχουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο υπέρ της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας. Δεύτερον, για την καινοτομία. Οι επενδύσεις σε νέες γεωργικές τεχνολογίες είναι κλειδί. Η έρευνα και η ανάπτυξη, υποδομές, η κατάρτιση, η μεταφορά τεχνογνωσίας είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και η ΚΑΠ πρέπει να έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής λέει ότι πρωταρχικός ρόλος ε, για τη Γεωργία είναι προμήθεια τροφίμων. Εμείς θεωρούμε ότι η παραγωγή τροφίμων και η ασφάλεια δεν επηρεάζεται από τους μη παραγωγούς. Eh, Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Επομένω, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τα μέλη του πάνελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, που πήραν το λόγο σήμερα και του ε, συναδέλφους μας. Και τώρα, Άλμπερ έχει τον λόγο για να ολοκληρώσει αυτή την τόσο σημαντική ημέρα. Ευχαριστώ Πάολο. Ευχαριστώ και όλους τους εμπειρογνώμονες ε, για τις τοποθετήσεις σας και ε, σε όλους τους συμμετέχοντες για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο Πάολο για τον τρόπο με τον οποίο διεύθυνε τη συνεδρίαση. Ε, για τα τρία θέματα, όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές, ε, σημείωσα πολλά ότι υπήρχε πλήρη συμφωνία ότι χρειαζόμαστε διατροφική ασφάλεια για μισό μισό δισεκατομμύριο ανθρώπων στην Ευρώπη ότι ε, αναφερθήκαμε στις θέσεις εργασίας και υπάρχουν ορισμένες ε, ε, παρανοήσεις διότι εγώ δεν μίλησα κατά των κοινωνικών πτυχών επίσης επιζητούμε να υπάρχει μία δίκαιη και σωστή κατανομή των πόρων αλλά δεν είπα και δεν προεξόφλησα τι θα πω στην έκθεσή μου. Μέχρι ότου τα γράψω έχω ο καιρό. Η μείωση της γραφειοκρατίας είναι κάτι που μας ενδιαφέρει αλλά ίσως θα πρέπει να μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη λέξη. Δεν θέλουμε να ε, πανεθνικοποιήσουμε την γεωργική πολιτική αλλά χρειαζόμαστε ε, μία αντιστάθμιση των μεγάλων διαφορών μεταξύ κρατών μελών και των ε, τοπικών και περιφερειακών αγορών που είναι πιο απρόμακρες και πρέπει να ρυθμιστούν από τις Βρυξέλλες. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά των κρακών μελών χωρίς να υπάρχει επανεθνικοποίηση. Όσον αφορά τα δημόσια αγαθά και τα τρόφιμα που παράγονται ε, πιστεύουμε ότι ένας γεωργός είναι πάντα γεωργός ασχέτως της μορφής της παραγωγής του. Ευχαριστώ για το σχόλιο για τους μικρούς γεωργούς για τους οποίους πρέπει να υπάρχει ένας ορισμός. Το ανώτατο όριο το πλαφόν θα παραμείνει πάντοτε αμφιλεγόμενο σημείο αλλά θα ήθελα να μου είχατε απαντήσει σχετικά με τον ε, διαχωρισμό των ε, περιβαλλοντολογικών μέτρων μεταξύ πρώτου και δευτέρου ε, πυλώνα γιατί εκεί έχω πρόβλημα. Εγώ δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό αλλά θα ήθελα μία, με ένα μέρος των πληρωμών να μετατεθούν από το πρώτο στο δεύτερο πυλώνα χωρίς συγχρηματοδότηση ε, για να μην ε, συγχέουμε τα μέτρα μεταξύ πρώτου και δευτέρου πυλώνα και να μην υπάρχει ε, και να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Θα είχαμε λιγότερα μέτρα αλλά μεγαλύτερη ευελιξία όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν ήδη στο δεύτερο πυλώνα και αν δεν υπάρχει συγχρηματοδότηση για τον γεωργό που είναι το πρόβλημα. Τέλος, όσον αφορά τα μέτρα για τις αγορές, θα ήθελα να περιοριστούν οι διακοιμάσεις των τιμών σχετικά με το Μιερκοσούρ. Ε, άκουσα ότι σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας απεφασίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναβάλει τις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική από ό,τι στην προηγούμενη θητή διότι πρέπει καταρχήν να συμφωνήσουμε στο επίπεδο του ΠΟΕ και να μην ε, ε, αποφασίζουμε μέσω διμερών ε, συμβάσεων. Όσον αφορά την έκθεση για τις μεταρρυθμίσεις στη Γεωργία, τι όφελος θα έχει να υπερψηφιστεί αν εντωμεταξύ έχουμε προεξοφλήσει και προκαταλάβει τα αποτελέσματα αποτελέσματα. Όσον αφορά την ε, ε, αστάθεια των τιμών, αντιλαμβάνουμε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αποθήκευση διότι ε, πώς θα αποφύγω την κερδοσκοπία εάν υπάρξει αύξηση τιμών και δεν έχω, δεν έχω απόθεμα. Όταν μιλάμε για 10 κιλά σιτηρά ανακατοικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ένα μικρό ποσό το οποίο θα πρέπει να υπάρχει ε, ε, αποθηκευμένο διότι δεν πρέπει όλα τα έξοδα να τα αφήνουμε μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία διότι τότε είμαστε δέσμοι της κερδοσκοπίας. Ε, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα λέγοντας ότι θα περιορίσουμε αφήσουμε απλώς τις τιμές προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πρέπει μέσω των μέτρων της αγοράς να μπορούμε να επεμβαίνουμε. Επίσης οι ενισχύσεις για τη γεωργία και ευχαριστώ που όλοι είπαν ότι οι ενισχύσεις πρέπει ε, να απευθύνονται στους καταναλωτές ή ε, στις σταθερές τιμές και αν η Ευρώπη ε, διαθέτει ένα 10% των πόρων για τη γεωργία υπάρχουν ε, ε, κεφάλαια τα οποία έχουν αποδοθεί με λιγότερο αποτέλεσμα σε άλλους τομείς και πρέπει να συνυπολογίσουμε και την κοινωνική σημασία. Όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, τους στόχους, τις προτεραιότητες στο στρατηγικό χώρο ο οποίος αναφέρθηκε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να διευκολύνουμε τις διαδικασίες κατά τρόπον ώστε να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη στην Ήπεθρο και αντιλαμβάνουμε ότι επειδή ήμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση πολιτικό σε πολλά χρόνια μέσω του δεύτερου πληλώνα υπήρξε μία κατανάλωση πόρων που δεν έδωσαν σωστά αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας την Ήπεθρο και ε, να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα θέματα και να τα συμπεριλάβουμε στις σκέψεις μας. Όπως ελέγχθηκε προηγουμένως ε, μετά από την ανακοίνωση του Επιτρόπου Τσόλος άκουσα πολλά, ε, ε, πολλά πολλές προτάσεις αλλά όπως λέγεται ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες και πρέπει να τον εξορίξουμε οπότε θα δούμε τι γίνεται και όταν υπάρχουν εκπρόσωποι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγώ πρέπει να πω στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εξέπληξε ότι ε, ε, όταν άκουσα τα ονόματα των 27 ε, επιτρόπων ότι ο Επίτροπος Γεωργίος ανεφέρθηκε στην 27η θέση αντί στη δεύτερη ή τρίτη που θα έπρεπε να έχει η θέση της Γεωργίας. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στην ακρόαση αυτή. Θα είμαστε σε επαφή. Ε, αρχές Φεβρουαρίου θα δώσω το έγγραφό μου για μετάφραση και θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ Άλμπερτ. Σας υπενθυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα την 1η Φεβρουαρίου στις 3. Ευχαριστώ σε όλους, όλους τους εμπειρογνώμονες. Ε, θα τα πούμε σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.